Are you sure? Yesterday I trouble. Good morning. Καλημέρα σας, είπα. Περιμέναμε μήπως έρθουν κι άλλοι, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Εχθές το απόγευμα θα θυμάστε ότι έγινε το πρώτο μέρος αυτής της ακρόασης για την διακυβέρνηση και αξιολόγηση του Σέγγεν. Στο πρώτο τμήμα ήρθε η Επίτροπος Μάλστρομ και ο Ιρλανδός Υπουργό Σάτερ καθώς και ακούσαμε τον εισηγητή Κάρλος Κουέλιο. Σήμερα στο δεύτερο τμήμα θα συζητήσουμε πώς έχει η τεχνολογία και θα συζητήσουμε μερικά εργαλεία στα οποία, επί των οποίων έχουμε συνομοθετήσει στο παρελθόν και τώρα θα θέλαμε να μάθουμε πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Σας θυμίζω όλους και όλες ότι οι ερωταπαντήσεις θα γίνουν μετά τις παρουσιάσεις από τους τέσσερις ομιλητές που έχουμε εδώ. Θα ακολουθήσουμε το πρόγραμμα όπως το γράφει. Αρχίζουμε λοιπόν με τον κύριο Τούντορατς που θα εκπροσωπήσει την Κομισιόν και θα μας μιλήσει για τις τελευταίες εξελίξεις ως προς το ΣΥΣ 2 αλλά και το DIS βέβαια και μετά θα ακούσουμε τους υπόλοιπους προσκεκλημένους μας που τους καλυσερίζουμε τον κύριο Γκάρκοφ που είναι διευθυντής της υπηρεσίας, ποιας υπηρεσίας τον κύριο Λάρκνερ, Λέκνερ μάλλον, Διευθυντή του Ιδρύματος για την Προστασία και Ασφάλεια των Πολιτών και τέλος και τον κύριο Μπέλσερ για το σχέδιο Fidelity. Πρώτα θα μας μιλήσει ο κύριος Τούντορακ της Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι. Σα ευχαριστώ επίσης για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας, της ακρόασης δηλαδή. Είναι όντως, ήταν όντως καιρός να δούμε πώς έχουν τα πράγματα και για το ΣΥΣ2. Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω τις λεπτομέρειες του ιστορικού για το ΣΥΣ2 γιατί τα έχετε δει, τα έχετε ζήσει Έχετε δει τις δυσκολίες του τα τελευταία δέκα χρόνια, καθυστερήσεις, αποτυχίες, υπερβάσεις του προϋπολογισμού και πολύ έντονες συζητήσεις στο Συμβούλιο και εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή σας. Η ιστορία αυτή λοιπόν ήταν, υπήρξε δύσκολη σήμερα. Μπορούμε να δούμε και να δείξουμε όπως βλέπετε στην οθόνη ότι το ΣΥΣ 2 θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 9η Απριλίου 2013. Είναι λοιπόν μεγάλο επίτευγμα αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας γιατί πιστέψατε στο ΣΥΣ 2 σε εποχή όπου οι άλλοι δεν πίστευαν στις δυνατότητες που έχει. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Κοέλιο που ήταν ίσως ο στεναρότερος υποστηρικτής του. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ κύριε Κοέλιο για την υποστήριξη και όσα κάνατε ώστε η 9η Απριλίου να καταστεί δυνατή. Θα σας αναφέρω πού βρισκόμαστε πρώτα γιατί είναι θέμα τεχνολογικών εξελίξεων και να σας εξηγήσω γιατί στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου συζητήθηκαν και άλλες καθυστερήσεις που οφείλονταν στα κράτη-μέλη και πώς μέσα σε τρεις μήνες καταφέραμε να, πούμε, να λέμε σήμερα ότι σε τόσο λίγο διάστημα, σε τρεις εβδομάδες θα αρχίσει να εφαρμόζεται το ΣΥΣ2. Η καθυστερήση ήταν σταθερό χαρακτηριστικό της ιστορίας του ΣΥΣ. Σε συνεργασία με τους τελικούς χρήστες και τα κράτη-μέλη καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που είχαν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο μερικά κράτη-μέλη στις δοκιμές τους και στις αρχές του έτους συμπληρώθηκαν όλες. Στα τέλη του Ιανουαρίου άρχισε το λεγόμενο Live Data Migration, δηλαδή φορτώσαμε στο σύστημα τα 46 εκατομμύρια στοιχεία που διαθέταμε χωρίς κανένα πρόβλημα και τις περασμένες δύο εβδομάδες τα κράτη-μέλη άρχισαν να φορτώνουν και τις δικά τους στοιχεία στο σύστημα. Και αυτό μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει συμπληρωθεί. Και όλα αυτά για να γίνει η μεταφορά, η αλλαγή στις την 9η Απριλίου. Οπότε και τα κράτη-μέλη θα ανάψουν το ΣΥΣ 2 και θα αρχίσουν να μπορούν να το χρησιμοποιούν άμεσα στη θέση του παλιού ΣΥΣ. Από την 9η Απριλίου λοιπόν και μετά, ίσως να το ξέρετε γιατί και χάρη σε εσά καταφέραμε το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας να διορθώσουμε νομικά τουλάχιστον τις τεχνικές διαδικασίες που αντιπροσωπεύουν τη μεταφορά των στοιχείων από το ένα σύστημα στο άλλο. Και πάλι λοιπόν σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας γιατί μας δώσατε ένα σαφές πλαίσιο για την μεταφορά και για το σβήσιμο του ΣΥΣ 1 και το άναμα του ΣΥΣ 2. Η ενδιάμεση περίοδος Κατά την ενδιάμεση περίοδο θα διατηρούνται ζωντανά και τα δύο συστήματα, ώστε αν κάποιο κράτος μέλος έχει πρόβλημα να μεταφέρει τη λειτουργία στο νέο σύστημα, να μπορεί να λειτουργήσει ακόμη το παλιό. Από τεχνικής απόψεως λοιπόν και από πλευρά της ετοιμότητας, αυτά προβλέπονται τις επόμενες εβδομάδες και είπαμε ότι την 9η Απριλίου γίνεται η επίσημη μεταφορά και μετά από ένα μήνα επιτήρησης στις 9 Μαΐου ξέρετε ποια σημασία έχει η ημερομηνία αυτή στις 9 Μαΐου λοιπόν το ΣΥΣ 2 θα είναι πλήρως λειτουργικό και θα είναι πια το μόνο σύστημα πληροφόρησης του χώρου Σέγγεν. Τώρα, ποια είναι τα ωφέλη του ΣΥΣ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα αναφέρω λεπτομερώς. Τα έχουμε πει ποια είναι. Καταρχήν η διακυβέρνηση, governance, είναι η μεγαλύτερη εξέλιξη σε σύγκριση με το ΣΥΣ 1. Το ΣΥΣ 2 θα είναι καθαρά ενωσιακό εργαλείο και πλήρως ενωσιακό. Επίσης ως προς την διαχείρισή του, η διαχείριση θα γίνεται από την υπηρεσία Ουλίσα. Ούτε γι' αυτό θα αναφέρω λεπτομέρειες γιατί ο κύριος Γκάλκοφ θα ακολουθήσει μετά και θα, σα... και θα σας τα πει ίσως και εκείνος πώς λειτουργεί δηλαδή αυτή η υπηρεσία για την καλύτερη διαχείριση των συστημάτων με μεγαλύτερη λογοδοσία. Πράγμα που είναι χρήσιμο όχι μόνο για τα θεσμικά όργανα εδώ αλλά και για τους πολίτες. Δεύτερον, το SIS2 είναι καλύτερη τεχνολογία. Αυτός είναι βέβαια ο κύριος λόγος για τον οποίο θελήσαμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί όλοι συμφωνούσαν ότι χρειαζόμασταν καλύτερη τεχνολογία από του sis 1 Δοκιμάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια και τελικά μπορούμε να διαχειριζόμαστε ε, μέχρι 100 εκατομμύρια δελτία. Η αποδοτικότητά του ξεπερνάει το ΣΥΣ 1 τουλάχιστον κατά 200% και τέλος το ΣΥΣ 2 έχει και νέες λειτουργίες δηλαδή δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούν οι διάφορες αιτήσει ή οι διάφορες, οι διάφορες προειδοποιήσεις να συνεννοούνται καλύτερα τα αστυνομικά σώματα μεταξύ τους και να συνδέονται οι πληροφορίες με άλλες πληροφορίες. Τέλος, είναι και καλύτερη προστασία για τους πολίτες, περισσότερες εγγυήσει. Γιατί καμιά φορά υπήρχαν προβλήματα για τους πολίτες όταν υπέβαλαν κάποιο αίτημα ή παράπονο. Τέλος, η προστασία των δεδομένων, το ΣΥΣ έχει αυξημένες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων, όχι μόνο με όρους governance, διότι ο επόπτης, ο ενωσιακός επόπτης, ε, θα, επιτηρητής θα γίνει ο κύριος υπεύθυνος για την ασφάλεια των δεδομένων του κεντρικού συστήματος, αλλά και γιατί θα λειτουργεί σε συνεργασία και με εθνικές αρχές για την προστασία των δεδομένων. Γενικά, το, η προστασία των δεδομένων του ΣΥΣ2 είναι πολύ μεγαλύτερη από του προηγούμενου συστήματος. Ας περάσω τώρα στο ΒΙΣ. Το ΒΙΣ είναι άλλο πράγμα. Λειτουργεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2011. και λειτουργεί από τότε χωρίς προβλήματα, χωρι... εξυπηρετώντας τα κράτη-μέλη μέχρι τώρα ήδη 2,5 εκατομμύρια θεωρήσεις έχουν αναλυθεί από κείνο σε 12 περιφέρειες ή χώρες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσουν τις 15. Μέχρι τώρα δεν έχει σημειωθεί κανένα πρόβλημα από τεχνολογικής απόψεως και το ίδιο το out θα χρειαστεί, χρειάζεται μερικούς μήνες ή και ένα-δυο χρόνια ανάλογα με την ετοιμότητα των, της προετοιμασίας που θα έχουν ορισμένες περιφέρειες ή χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία. Ούτως ή άλλως η υπηρεσία που ασχολείται ήδη με την λειτουργήση του ΒΙΣ ήδη προσπαθεί να το βελτιώσει τεχνολογικά για να στηρίζει πλήρως το σύνολο της διαδικασίας. Η τεχνολογία δηλαδή του ΒΙΣ θα στηρίζει πλήρως τους πολιτικούς στόχους που του έχουν τεθεί. Ευχαριστούμε κύριε Τούντορακ. Να προχωρήσουμε τώρα στον κύριο Κρουμ Κάρκοφ, ο οποίος είναι εκτελεστικός ε, διευθυντής της επιχειρησιακής ε, διαχείρισης της υπηρεσίας για την υπηρεσιακή διαχείριση για τον ε, συστήματα πληροφορικής στον τομέα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Ακούσουμε την άποψή σας σχετικά με την κατάσταση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα να περιβρίσκουμε εδώ και να σας ενημερώσω σχετικά με την πρόοδο του Ιουλίσα. Εδώ και λίγους, μόνο, και λίγους μόνους μήνες ε, υπάρχει. Άρχισε η υπηρεσία να λειτουργεί την 1η Δεκεμβρίου, ομαλά, λόγω της ε, υποστήριξης που είχε από τα κράτη-μέλη και κυρίως από τα κράτη-μέλη όπου βρίσκεται η έδρα της ε, υπηρεσίας του οργανισμού και η Κομισιόν ε, προετοιμάστηκε πολύ καλά εκ των προτέρων. Έχουμε δύο προτεραιότητες. Καταρχήν είναι να συνεχίσουμε την πρόσληψη του προσωπικού έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε το καθήκον μας και κατόπιν να ξεκινήσουμε την ε, μεταφορά καθηκόντων σε σχέση με την επιχειρησιακή διαχείριση των συστημάτων. Σε ό,τι αφορά την πρόσληψη προσωπικού, να σας πω ότι η υπηρεσία ε, προσλαμβάνει τώρα προσωπικό. Έχουμε σεβαστεί το σχέδιο για το 2012. Τώρα έχουμε 81 άτομα στο Στρασβούργο και στο Τάλιν και επίσης έχουμε και 32 κοινές, ε, κοινές θέσεις. Συνεχίζονται οι διαγωνισμοί και στο τέλος του έτους αναμένουμε ότι θα μπορέσουμε να σεβαστούμε και το σχέδιο προσωπικού για το 2013 θα έχουμε δηλαδή άτομα, 120 άτομα προσωπικό. Επίσης ε, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων και ήδη έχουμε έναν υπεύθυνο προστασίας ε, των δεδομένων και έναν ε, υπεύθυνο που ε, διασφαλίζει ότι ξεκινούν ομαλά οι επιχειρήσεις ε, από οικονομική σκοπιά. Σε ό,τι αφορά την μεταφορά ευθυνών, τη διαβίβαση των ευθυνών από την πρώτη μέρα ύπαρξης του οργανισμού, συνεργαστήκαμε με τις Γαλλικές Αρχές και με την Κομισιόν και συστήσαμε ένα κοινό σχέδιο υπηρεσίας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η διαβίβαση ευθυνών θα γίνει ομαλά και γέρος και δεύτερον να διασφαλίσουμε την ένταξη ε, του προσωπικού της γαλλικής ομάδας που μέχρι την 1η Δεκεμβρίου ήταν ε, υπεύθυνα για την επιχειρησία και διαχείριση των συστημάτων. Επίσης, χαίρομαι να σας ενημερώσω ότι σήμερα ε, προχωρούμε σύμφωνα με το πρόγραμμα στην εφαρμογή του σχεδίου μετάβασης και ε, ελέγχουμε πλήρως το VIS. Επίσης, ε, η υπηρεσία εργάζεται με έναν ανάδοχο για θέματα συντήρησης, για την επιχειρησιακή συντήρηση, αλλά και για την εξέλιξη του συστήματος VIS για να αντιμετωπίσουμε τις καθολικές ανάγκες αλλά και τις ανάγκες που θα εντοπίσουν τα κράτη-μέλη σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος. Σε ό,τι αφορά τη Eurodac, αυτή τη στιγμή η μεταφορά των ευθυνών της Eurodac ε, προχωράει Πολλές από τις σχεδιασμένες δραστηριότητες έχουν ήδη υλοποιηθεί σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση γνώσεων από την ομάδα της Κομισιόν στην ομάδα της υπηρεσίας και μέχρι τα τέλη Μαΐου. Η υπηρεσία θα ελέγχει πλήρως και τη Eurodac. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, αν και ο οργανισμός θα αναλάβει τις ευθύνες για την επιχειρησιακή ευθύνη του ε, ΣΥΣ μετά τα τέλη Μαΐου, από τις αρχές αυτού του έτους, ο οργανισμός ήδη συνεισφέρει και συμμετέχει στι εναπομείνε δραστηριότητε για τη μετάπτωση των δεδομένων και σε ό,τι αφορά και τις προετοιμασίε για την μετάβαση που θα γίνει, για το switch over που θα γίνει στα τέλη Απριλίου. Έτσι λοιπόν από τις 9 Απριλίου βασικά θα αρχίσουμε να ε, παράγουμε αποτελέσματα για το SIS, για το SIS και αυτό θα αποτελέσει μια καλή ενέργεια για να αναλάβουμε την ε, πλήρη ευθύνη μετά τις 9 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες για φέτος, ε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ευρύτερη εικόνα, γιατί μέχρι τώρα αναφέρθηκα σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τη διαχείριση της Νοτισολά. Εμείς έχουμε και ένα πρόγραμμα εργασίας για το 2013 και νομίζω είναι σημαντικό αυτή η Επιτροπή να έχει και μια εικόνα για τις πλήρες δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για την υπηρεσία φέτος. Για φέτος ε, έχουμε τέσσερις προτεραιότητες. Η μια αφορά το να υλοποιήσουμε τα κύρια καθήκοντα, έτσι όπως προβλέπεται από τον κανονισμό σύστασή μας. Δεύτερη προτεραιότητα, να οικοδομήσουμε την οργάνωση της υπηρεσίας με την πρόσληψη των κατάλληλων ατόμων. Τρίτον, κάτι που προέρχεται κατευθείαν από τις διατάξεις του κανονισμού. Θα προετοιμάσουμε το έδαφος ε, για να μετατραπούμε σε ένα κέντρο αριστείας τα επόμενα έτη και τέλος, θα δημιουργήσει υπηρεσία σχέσεις με τους εταίρους, εσωτερικούς εταίρους, δηλαδή με άλλες υπηρεσίες, άλλους οργανισμούς, αλλά και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, τα κράτη-μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη εδώ στις Βρυξέλλες, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θέλω να σας αναφέρω κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για τα δικά μου καθήκοντα έχουμε ως κυρία προτεραιότητα τη διαχείριση των συστημάτων μαζί με την ασφάλεια και τα, η προστασία των δεδομένων, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι γίνεται σωστή χρήση των δεδομένων και τα φυλάσσουμε σωστά. Επίσης, ε, θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε ορισμένα στρατηγικά σχέδια της εξελίξης του ΔΙΣ, όπως ανέφερα, αλλά θα μεταφέρει και το σύστημα Eurodac από το Λουξεμβούργο στο Στρασβούργο και μόλις η αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac θετηθεί θα αρχίσουμε τις εργασίες μας. Επίσης θα υποστηρίξουμε προδραστικά τα κράτη-μέλη που πρόκειται να μπουν στα συστήματα που θα ελέγχει η υπηρεσία σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση της οργάνωσης. Η κύρια προτεραιότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πρόσληψης γιατί το προσωπικό θα είναι ζωτική σημασία για φέτος αλλά και για του χρόνου προκειμένου ο οργανισμός να αρχίσει να λειτουργεί. Επίσης, θυμάμαι ότι η πρώτη φορά που ήρθα να μιλήσω σε αυτή την επιτροπή με προειδοποίησαν φιλικά ότι ε, μια διαίρεση του οργανισμού μπορεί να δημιουργήσει κάποιες ε, προκλήσεις. Το γνωρίζουμε αυτό και η Πρισσίδη έχει ήδη καθορισμένη την αποστολή της, η οποία αντικατοπτρίζεται στις επιχειρήσεις μας και υπάρχει στέρεη βάση για να αναπτύξουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση. Επίσης, θέλουμε να πετύχουμε οικονομική ανεξαρτησία αργότερα φέτος, μέχρι τα τέλη Μαΐου, και να δώσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, να παράσχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο μια στρατηγική για το 2014-2020 γιατί χρειάζεται μια διεύθυνση για την υπηρεσία βάσει τη στρατηγική που ελπίζω να υιοθετήσουμε μέχρι τα τέλη του 2013. Σε ό,τι αφορά τώρα το κέντρο αριστείας. Φέτο ε, θα επικεντρωθούμε στο να αναπτύξουμε ένα ε, πλήρε πλαίσιο διακυβέρνηση, αλλά και να αναθεωρήσουμε και να εφαρμόσουμε τις βελτιώσεις ε, των υφιστάμενων διαδικασιών ε, που θα μας επιτρέψουν να έχουμε πιο αποδοτικές επιχειρήσεις όπως το κόστος ε, και να βελτιώσουμε το συνολική αποτελεσματικότητα του κόστους ε, της υπηρεσίας. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω σε ό,τι αφορά το πλαίσιο διακυβέρνησης. Αυτό έχει καθοριστεί και το Συμβούλιο άρχισε ήδη να εκπονεί ένα χάρτη πορείας για την εφαρμογή του αυτή θα είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες μας φέτος, αλλά και τα επόμενα έτη, γιατί η εφαρμογή υγιούς διακυβέρνησης δεν θα γίνει μέσα σε ένα έτος. Και τέλος, ως προς τις προτεραιότητες, από τις πρώτες μέρες η Βηρησία άρχισε να αναπτύσσει τις σχέσεις της ε, με τους εταίρους και τους stakeholders, την ενδιαφερόμενα μέρη, έχει εξαιρετική σχέση με τους εκπροσώπους των κρατών μελών και με τις συμβουλευτικές ομάδες ως ε, μέρος ε, της δομής διακυβέρνησης και όλοι μαζί αντιμετωπίζουμε τα διάφορα επιχειρησιακά στρατηγικά θέματα που έχουν να κάνουν ε, με την εξέλιξη των συστημάτων ή με την προετοιμασία επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα η υπηρεσία έχει αναπτύξει πολύ στενή σχέση και σε εκτελεστικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο με άλλες ε, υπηρεσίες που έχουν στην πολιτική μας, καταρχήν με τη Europol, με τη Frontex, με το EASO, με τη SEPOL και Ήδη έχουμε το πρώτο μνημόνιο κατανόηση με τη ΣΕΠΟΛ. Έχουμε συμφωνήσει από αυτού για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένε ανάγκε που προέρχονται από τον κανονισμό ίδρυση της υπηρεσίας. Αυτή η εταιρική σχέση θα μεγεθυνθεί κατά τη διάρκεια του έτους ε, και το ίδιο ισχύει και για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Έχουμε διασφαλίσει ότι πάντοτε θα λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες και τις απόψεις των κρατών μελών σε σχέση με την ανάπτυξη των συστημάτων και των επιχειρήσεων γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι ο κύριος σκοπός, δηλαδή να προσδώσουμε αξία για τους stakeholders βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Φυσικά, τους πρώτους μήνες επίσης αντιμετωπίσαμε πολλά ζητήματα, όπως κάθε νέος οργανισμός, όμως ε, τα κύρια που αντιμετωπίζουμε νομίζω επιτυχώς μέχρι τώρα και πάλι αφορούν το προσωπικό, αυξάνονται επιχειρήσεις, μεγαλώνουν οι ευθύνες, τα καθήκοντα που αν λοιπόν, στην υπηρεσία πιθανότατα θα μεγεθούν του επόμενου μήνε και αυτό θα την πολύ μεγάλη πίεση στο σημερινό προσωπικό αλλά και στην υπηρεσία για να μπορέσει να εξελιχθεί πολύ νωρίτερα από τα τέλη του έτους. Επίσης, η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε φέτος αλλά και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια είναι να αναπτύξουμε τις στρατικές μας ικανότητες ως προς το σχεδιασμό και την έρευνα ε, και την αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων σε ένα δύσκολο οικονομικό κλίμα που πολλές φορές μπορεί να μας εμποδίζει να προχωράμε όσο γρήγορα θα θέλαμε. Και τέλος, Ένα άλλο ζήτημα μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στο Στρασβούργο είναι οι συνθήκες εργασίας εκεί. Παρόλο που χρησιμοποιείται ο χώρος αυτή τη στιγμή από την υπηρεσία, δεν αρκεί η χωρητικότητα για το προσωπικό που έχουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις στρατηγικές ανάγκες της υπηρεσίας και νομίζω ότι αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί τους επόμενους μήνες σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να κλείσω. Η έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας ήταν επιτυχής. Αυτή τη στιγμή επιταχύνουμε τις εργασίες μας όπως έχουμε σχεδιάσει. Το πρόγραμμα εργασίας ε, επίσης προχωρά σύμφωνα με το σχεδιασμό και να τονίσω ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα και η επιτυχή επίλυσή του οφείλεται στην επιτυχή συνεργασία που αναπτύξαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις Γαλλικές Αρχές, κυρίως στο Στρασβούργο, αλλά και με τα άλλα κράτη-μέλη που φιλοξενούν την ε, υπηρεσία και όλα τα άλλα κράτη-μέλη που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα περνάμε σε ένα άλλο θέμα, στα βιομετρικά διαβατήρια. Θα μας μιλήσει ο κύριος Λέχνερ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Ιδρύματος για την ασφάλεια των πολιτών του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου. Θα μας παρουσιάσει κάποια επαγγελματικά πορίσματα σε ό,τι αφορά το όριο ηλικία για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι. Να σας παρουσιάσω εδώ μια προκαταρκτική παρουσίαση των πορισμάτων μιας μελέτης που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, την οποία ε, διεξήγε το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο το ερευνητικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όποιοι δεν γνωρίζουν το κοινό ερευνητικό κέντρο, να σας πω ότι πρόκειται για πλήρη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μοναδικό μέρος όπου γίνεται κατευθείαν έρευνα. Δεν ανατίθεται εξωτερικά, γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέτοια έρευνα. Το κοινό ερευνητικό κέντρο ε, έλαβε λοιπόν εντολή να διεξάγει αυτή την εντολή από τη Γενική Διεύθυνση Home Δίνουμε λοιπόν συμβουλές σε ό,τι αφορά τεχνολογικά και επιστημονικά ζητήματα. στόχος της μελέτης ήταν σαφής από την αρχή, από το έτος 2008 γίνεται συζητήσεις για τα δακτυλικά αποτυπώματα ανηλίκων στο πλαίσιο των συστημάτων που αναφέρθηκαν. Ετέθηκε το ερώτημα κατά πόσον υπάρχει κάποιο ελάχιστο όριο ηλικιακό από το οποίο μπορεί κανείς να πάρει δακτυλικά αποτυπώματα. Και φυσικά όλοι πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν τα παίρνουμε πλέον με μελάνι, αλλά ψηφιακά. Και εδώ λοιπόν τίθενται τεχνολογικά ζητήματα και επίσης η αναγνώριση, ο εντοπισμός των αποτυπωμάτων γίνεται ηλεκτρονικά. Τα θέματα λοιπόν τα οποία εξέτασε η μελέτη ήταν τα εξή. Καταρχά το θέμα της ανάπτυξης. Φυσικά τα παιδιά αναπτύσσονται αναπτύσσονται και τα δάχτυλά τους και μαζί με αυτά και τα αποτυπώματα. Το ερώτημα λοιπόν είναι κατά πόσον τα μεγαλύτερα αποτυπώματα, καθώς μεγαλώνει ένα παιδί, μπορούν να αναγνωριστούν ακόμα μετά από κάποια χρόνια. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσον οι αλγόριθμοι και η τεχνολογία μπορούν να αναγνωρίσουν παλαιότερα τα αποτυπώματα. Δεν είναι θεωρητικό το ζήτημα. Δεύτερο ερώτημα. Αν είναι πιο μικρό το δακτυλικό αποτύπωμα, τα χαρακτηριστικά καλύπτουν μικρότερη επιφάνεια. Είναι πιο πυκνά. σε ό,τι αφορά τις κανονικές ε, γραμμές των αποτυπωμάτων. Άρα λοιπόν είναι η ανάλυση της εικόνας επαρκής. Αυτά τα δύο ερωτήματα αρχίσαμε να ερευνούμε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε πρόκειται για κάτι περίεργο. Από ό,τι καταλαβαίνετε πρέπει κανείς ε, για να κάνει αυτή την έρευνα να έχει τακτιλικά αποτυπώματα ενός ατόμου με κάποια χρονική απόσταση. Δεν φτάνει δηλαδή να πάρουμε αποτυπώματα μία ηλικία από ένα παιδί. Θα πρέπει το ίδιο παιδί μετά από κάποια χρόνια να του ξαναζητήσουμε να πάρουμε τα αποτυπώματά του από το ίδιο δάκτυλο, από το ίδιο παιδί. Και καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχαν τόσο πολλά δεδομένα διαθέσιμα Τουλάχιστον δύο φορές με κάποια χρονική απόσταση πρέπει να πάρουμε αποτύπωμα. Και όταν κανείς ξεκινάει από την αρχή μια τέτοια μελέτη, ε, αν για παράδειγμα πρέπει κανείς να δει πώς αναπτύσσονται τα αποτυπώματα μετά από τρία χρόνια, θα πρέπει και η ίδια η μελέτη να διεξαχθεί σε τέτοια χρονική περίοδο. Είμαστε λοιπόν πολύ ευγνώμονες στην πορτογαλική κυβέρνηση που μας έδωσε ανώνυμα αποτυπώματα παιδιών. Δεν είχαμε καθόλου ονόματα, μόνο τα αποτυπώματα. Δεν θέλω να μπω σε μια φιλοσοφική συζήτηση για την ανωνυμοποίηση. Απλά αναφέρω ότι ήταν η ευγενική προσφορά της πορτογαλικής κυβέρνησης τα αποτυπώματα αυτά. Και μεταβιβάστηκαν στο κοινό ερευνητικό κέντρο με τι υψηλότερε προδιαγραφέ ασφαλεία. τα μετέφερα εγώ τα στοιχεία αυτά στον χαρτοφύλακά μου από την Πορτογαλία στο αεροδρόμιο. Ήταν λοιπόν πολύ σαφή η όρη τη σύμβαση και έγιναν σεβαστοί. Τα χαρακτηριστικά τα οποία εξετάσαμε, εξετάσαμε αποτυπώματα 1600 παιδιών. Είχαμε πιο πολλά αποτυπώματα, δύο του αριστερού και του δεξιού δίκτυ, τα είχαμε σκανάρει ηλεκτρονικά δύο φορές με διαφορά χρονική δύο έως το 4,5 έτη. Η μέγιστη χρονική απόσταση ήταν 4,5 χρόνια και η κάλυψη ηλικιακή των παιδιών ήταν από 0 ε, έως 11 χρονών. Ε, χρησιμοποίησαμε τρεις αλγόριθμους. Βάσει τεχνολογικών αλγορίθμων λοιπόν μπορέσαμε να τις εξετάξουμε, αλλά δεν ε, άνοιξαμε τους αλγορίθμους αυτούς. Ήταν ένα μαύρο κυβότιο αν θέλετε. Μπήκε λοιπόν ε, το αποτύπωμα, μετά βγήκε ο αλγόριθμος και μετά με βάση αυτόν τον αλγόριθμο εξετάσαμε το κατά πόσον ε, υπήρχε ποσοστία αναγνώριση. Έτσι λοιπόν δομούνται τεχνικώς πώς οι αργόριθμοι και το ποσοστό ταυτοποίηση ήταν το ποσοστό το οποίο λάβαμε υπόψη για να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαν να γίνουν αναγνωρίσιμα τα αποτυπώματα. Και τώρα λοιπόν επανερχόμαστε στα δύο ερωτήματα που είχαμε θέσει στην αρχή. Τι γίνεται με, το, με την ανάπτυξη, το μέγεθος και με την πυκνότητα του αποτυπώματος. Και διαπιστώσαμε έκπληκτη ότι το θέμα της ανάπτυξης, του μεγέθους, δεν φαίνεται ότι αποτελεί θέμα. Τα αποτυπώματα τα οποία ε, μελετήσαμε, ναι, μεν μεγάλωσαν, δεν άλλαξαν όμως με την παράδοση του χρόνου. Αυτό ίσχυε ακόμα και με τα αποτυπώματα που είχαν τη μεγαλύτερη χρονική απόσταση, 4,5 χρόνια. Δεν υπήρξε σημαντική αλλαγή. Αυτό είναι αρκετά καλό ως πόρισμα. Άρα υποθέτουμε βάσει του γεγονότος ότι η ανάπτυξη γίνεται με κανονικό ρυθμό, φαίνεται ότι διατηρούνται τα χαρακτηριστικά. Όταν δηλαδή το δάχτυλο έχει διπλασιαστεί, οι αλγόριθμοι φαίνεται ότι λειτουργούν για να γίνει αναγνώριση. Δηλαδή ένα μικρό αποτύπωμα το οποίο μεγαλώνει μετά από κάποια χρονική διάρκεια μπορεί και πάλι να εντοπιστεί, να αναγνωριστεί. Αυτό ήταν ε, κάτι που μας προκάλεσε έκπληξη, γιατί είχε ανακύψει το ερώτημα αυτό και στο παρελθόν, αλλά ποτέ δεν είχε εξεταστεί. Δεύτερο προκαταρτικό πόρισμα, προκαταρτικό τονίζω, είναι ότι και το μέγεθος δεν φαίνεται να αποτελεί ζήτημα. Κοιτάξαμε λοιπόν θέματα πυκνότητας και τα, τις 500 ε, τελείες ανά ίντσα, DPI, είναι ένα τεχνικό χαρακτηριστικό αυτό για την ανάλυση του αποτυπώματος. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ότι και πάλι με τον αλγόριθμο μπορεί να γίνει αναγνώριση. Αν πρόκειται όμως για μικρότερα αποτυπώματα από το αρχικό και πάλι μπορεί να γίνει αναγνώριση. Άρα τεχνικά οι 500, τα 500 DPI φαίνεται ότι αποτελούν ένα σταθερό μέτρο για την αναγνώριση ακόμα και μικρότερων αποτυπωμάτων. Άρα τα πορίσματα της ε, έρευνας είναι αρκετά θετικά. Κοιτώντα όμως τα τεχνικά πρότυπα, διαπιστώσαμε και κάτι άλλο. Το εξή. Η ποιότητα είναι πάρα πολύ σημαντική και στο στα στοιχεία που μας έδωσαν οι πορτογαλικές αρχές, διαπιστώσαμε ότι η ποιότητα ήταν κάτι το οποίο αυξανόταν με την ποιότητα. Άρα, είναι πάρα πολύ καθοριστική η ποιότητα της καταχώρησης. Όταν παίρνει κανείς αποτυπώματα και καταχωρίζει τα παιδιά, θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία των πρακτικών. Και μπορεί να χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί διαπιστώσαμε ότι τα αποτυπώματα των νεαρών παιδιών είχαν πολύ διαφορετική ποιότητα. Αυτό δεν λέει, δεν σημαίνει ότι ήταν κακή η ποιότητα απαραίτητα. Υπήρχαν αποτυπώματα με πολύ καλή ποιότητα μικρών παιδιών. Άρα αυτό καταδεικνύει ότι η ποιότητα έχει να κάνει με τη διαδικασία λήψης των αποτυπωμάτων. Και για παράδειγμα μπορεί το δάχτυλο να είναι στεγνό αλλά να έχει κάποια επικάλυψη ζάχαρης, για παράδειγμα, το οποίο δεν φαίνεται παρά μόνο στην ψηφιακή μορφή της λήψης του αποτυπώματος. Άρα η ποιότητα γενικά χειροτέρευε όσο πιο μικρά ήταν τα παιδιά. Από πλευράς λοιπόν της μελέτης μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι τα δάκτυλα των μικρών παιδιών πρέπει να τα προσέχουμε πιο πολύ κατά την διαδικασία καταχώρηση. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε αποτυπώματα, γιατί είδαμε πολύ καλή ποιότητα σε πολύ μικρά παιδιά, αλλά τη διαδικασία που ακολουθείται φαίνεται ότι είναι πιο σημαντική. Αυτά λοιπόν, συνοπτικά. που καταλήγουν στο πόρισμα ότι υπάρχει αναγνώριση για αποτυπώματα με χρονική απόσταση 4,5 ετών. Αυτό δεν είναι δεσμευτικό μπορεί να περιλαμβάνει και μικρότερες ε, χρονικές αποστάσεις. Ενδεχομένω να μπορούν να καλυφθούν και μεγάλες χρονικές αποστάσεις. Το μικρότερο μέγεθος των αποτυπωμάτων των παιδιών τεχνικά δεν φαίνεται να επηρεάζει σε αυτή την ανάλυση. Η ποιότητα δε των αποτυπωμάτων είναι καθοριστική, αλλά αυτό δεν ισχύει για τα παιδιά μόνο, ισχύει για όλα τα συστήματα λήψης αποτυπωμάτων. Χρειάζεται υψηλή ποιότητα για την αναγνωρισιμότητα. Πάντα λοιπόν είναι καθοριστικός παράγοντας η ποιότητα, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί τα παιδιά βάζουν τα δάχτυλα στο στόμα και γενικά ενδεχομένω να είναι πιο βρώμικα τα δάχτυλά τους από αυτά των ενηλίκων. Προκαταρτικά λοιπόν πορίσματα για να επανέλθουμε στα αρχικά ερωτήματα. Η ελάχιστη ηλικία δεν αποτελεί προαπαιτούμενο. Θα μπορούσαμε να πάρουμε αποτυπώματα και από παιδιά κάτω του έτους και πάλι θα ήταν τεχνικά άρτια τα αποτυπώματα για την αναγνώριση μετά από πέντε χρόνια, ίσως και μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η διαδικασία λήψης των αποτυπωμάτων θα είναι πάρα πολύ σημαντική, το είπα. Και επί της αρχής, αν ε, θέλαμε να ορίσουμε ελάχιστη ηλικία, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η λήψη των αποτυπωμάτων γίνεται με σωστό τρόπο. Και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε πραγματικά να ελαχιστοποιήσουμε την ε, ηλικία λήψη αποτυπωμάτων. Αυτά λοιπόν είναι τα πρωταρχικά πορίσματα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Η μελέτη έγινε μετά από εντόλη της Γενικής Διεύθυνσης HOME. Θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι Βρισκόμαστε σε φάση διατύπωσης της έκθεσης. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω τα προκαταρτικά αυτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και τώρα θα περάσουμε στο τέταρτο ομιλητή, ο οποίος ε, βρίσκεται σε αυτή την πλευρά του το Προεδρείο ο κύριος Μπέλτσερ, ο οποίος θα παρουσιάσει το Project Fidelity. Να σας ανακοινώσω ότι... Αν και... Αν και υπάρχει η παρουσίαση στα α, αγγλικά, η παρουσίαση θα γίνει στα Ολλανδικά. Άρα όσοι δεν καταλαβαίνετε Ολλανδικά, παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας. Γεια σας, ε, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για το γεγονός ότι παρουσιάζω ένα τμήμα του Project Fidelity. Το Fidelity ε, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2012 έως 2016 και πρόκειται για σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Για να σας δώσω μία μικρή παρουσίαση για το Fidelity, βασιζόμαστε στον έλεγχο των e-passports, των ηλεκτρονικών ε, διαβατηρίων, από την αίτηση μέχρι και τη χρήση των διαβατηρίων σε αυτοματοποιημένες συνολικές συναλλαγές. Το ηλεκτρονικό διαβατήριο δεν είναι τόσο παλιό μετά τις επιθέσεις της 11 η Σεπτεμβρίου του 2001 ε, τέθηκαν σε γρηγορότερη εφαρμογή. Ξεκινήσαμε, ο ΙΚΑΟ ξεκίνησε να γράφει προδιαγραφές ε, για διαβατήρια με βιομετρικά δεδομένα του κατόχου. Αυτές οι προδιαγραφές το 2004 ολοκληρώθηκαν και από το 2005 και μετά εκδόθηκαν και τα πρώτα βιομετρικά ε, διαβατήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο με αποτυπώματα και με φωτογραφία. Και αυτά, αυτές οι συστάσεις του ΙΚΑΟ ε, έληφθησαν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλήφθησαν στον κανονισμό για τα, ταξιδιωτικά έγγραφα και ασφαλώς και για τις θεωρήσεις. Κοιτώντα τις διαφορές μεταξύ διαβατηρίων και εγγράφων πηγής, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Διαπιστώνουμε καταρχάς ότι για τα διαβατήρια ισχύουν διάφορες νομοθεσίες και διάφοροι κανονισμοί από την από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν διεθνεί συμβάσει. όπου συμφωνήσαμε ότι αν μια χώρα Α εκδίδει ένα νέο διαβατήριο θα πρέπει να μας διαθέτει στη χώρα Β ένα δείγμα για να ξέρουμε τι κυκλοφορεί. Ο αριθμό των διαβατηρίων που κυκλοφορεί στο, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι περίπου 3.000, άρα είναι περιορισμένο αρκετά ο ρυθμός και οι ελεγκτέ μπορούν να τα ελέγχουν από διάφορα συστήματα. Υπάρχει το σύστημα Φάντο στην Ευρώπη, υπάρχει και το ISO και το Ellison. Όλα αυτά είναι συστήματα επαλήθευση για να ελεγχθεί αν ένα διαβατήριο είναι πραγματικό, αυθεντικό πρωτότυπο και το πλεονέκτημα των ταξιδιωτικών εγγράφων είναι ότι έχουν πάρα πολλά συστήματα και σχέδια επαλήθευση. Κοιτώντας λοιπόν τα, τα άλλα στοιχεία, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, ε, διεθνείς προδιαγραφές, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα έγγραφα πηγής, ε, σε ό,τι αφορά το Ολλανδικό, το Πορτογαλικό, το Αγγλικό έγγραφο πηγής. Ε. Ο αριθμός τέτοιων εγγράφων που κυκλοφορούν είναι άγνωστος. Κάναμε μία παρουσίαση στις ΕΠΑ πρόσφατα και είπαμε τότε ότι ενδεχομένως δεν είναι χιλιάδες αυτά τα ε, τα, έγγραφα πηγής που κυκλοφορούν. Μπορεί να είναι και 8.000. Δεν ξέρουμε όμως ε, τι ακριβώς κυκλοφορείς. Δεν υπάρχουν ε, ουσιαστικά συστήματα για τα έγγραφα πηγής. Δεν υπάρχουν και τέτοια χαρακτηριστικά ε, επαλήθευσης στην Ευρώπη έχουμε ελάχιστα πρότυπα για τα ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά έγγραφα. Έχουμε ένα εναρμονισμένο στίκερ και ένα εναρμονισμένο ε, έγγραφο παραμονής για υπηκόους τρίτων χωρών. Και σε ό,τι αφορά το υλικό, τις ε, τεχνικές ε, εκτύπωσης, τις ασφάλειες, τις τεχνολογίες επαλήθευσης υπάρχουν ενιαίοι κανόνες. Άρα υπάρχει προστασία από τέτοια έγγραφα πλαστά. Μπορούμε να εμπιστευόμαστε όμως γενικά τα διαβατήρια, γιατί όταν παρουσιάζει κανείς ένα διαβατήριο υπάρχει πάντα σύνδεση μεταξύ διαβατηρίου και των βιομητρικών στοιχείων του κατόχου, αλλά πρόκειται για τη σωστή ταυτοποίηση, γιατί συχνά διαπιστώνουμε ότι δίδονται έγγραφα με πλαστή ταυτότητα. Και στη Γαλλία φαίνεται ότι υπήρξε πρόβλημα μεγάλο με 500 τέτοια διαβατήρια. Να σας πω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά διαβατήρια, αλλά δεν αφορά μόνο τη Γαλλία, είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε κάποιο βαθμό. Τώρα, η η αλυσίδα ταυτοποίηση. Ξεκινάμε από την καταχώρηση κατά τη γέννηση και μετά χρησιμοποιούνται αυτέ οι ταυτοποιήσει σε διάφορα βήματα. Σε αυτό το πλαίσιο θα, θα κοιτάξουμε βασικά θέματα καταχώρησης και της έκδοσης της πράξη ε, πράξης γέννησης. Ένα σημαντικό ερώτημα το οποίο θα πρέπει να θέσουμε είναι το εξής γιατί έχουμε, δίνουμε τόσο πολύ μεγάλη προσοχή για διαβατήρια, ταυτότητες, θεωρήσεις κτλ. δημιουργώντας νομοθεσία και έχουμε, δίνουμε τόσο λίγη σημασία για τέτοια ε, έγγραφα πηγής Όλες οι χώρες λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτά τα έγγραφα πηγής ε, χρησιμοποιούν ό,τι θέλουν ουσιαστικά. Δεν υπάρχει κοινός μορφότυπος, δεν υπάρχει κοινό περιεχόμενο. Και δεν υπάρχουν ε, ε, ασφαλείας, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά αυτά τα έγγραφα καταχώρησης. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τα οι δικλείδε ασφαλείας, όπως για παράδειγμα δατογραφήματα. κάποια ειδικά χρώματα, κάποιες ειδικές ε, τεχνολογίες εκτύπωσης. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται πολύ περιορισμένα. Και έτσι λοιπόν είναι μεγάλη η δυνατότητα και μεγάλη η ποικιλία μορφών παραχάραξης και αυτό που σας είπα δεν δημιουργεί προβλήματα μόνο στην χώρα έκδοσης αλλά και στην χώρα Υποβολή των εγγράφων αυτών. Να σας αναφέρω την γαλλική περίπτωση, όπου πολλά ηλεκτρονικά διαβατήρια εκδόθηκαν. Στην ε, Ολλανδία έχουμε πάνω από χίλια άτομα που έχουν κανονικά νόμιμα ηλεκτρονικά διαβατήρια, τα οποία όμως έχουν εκδοθεί βάση πλαστού εγγράφου καταχώρησης. Άρα, με ένα τέτοιο τρίκ, κόλπο, μπορεί κανείς νόμιμα να διαμένει σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε μόνο στην Ευρώπη. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε παγκόσμιο επίπεδο ψάχνουμε λύσει στα πλαίσια του ΙΚΑΟ, που είναι ο οργανισμό που είναι υπεύθυνο στην έκδοση προδιαγραφών για τα διαβατήρια. Εδώ και πέντε χρόνια συζητάμε τι μπορούμε να κάνουμε για την καλύτερη ε, ασφάλιση αυτών των εγγράφων πηγή, των εγγράφων καταχώρησης που χρησιμοποιούνται για την έκδοση διαβατηρίων. Μόνο ο ΙΚΑΟ πρέπει να σας πούμε ότι δεν έχει αρμοδιότητα για να εκδώσει σχετικές προδιαγραφές. Η Ιντερπολ ε, κάνει μια αιτήσια συνέλευση κάθε χρόνο και συζητιέται το θέμα της ε, κατάχρησης τέτοιων εγγράφων και στα πλαίσια της Ιντρεπό, λοιπόν, θέλουν να εκδώσουν ένα ψήφισμα για την καλύτερη ασφάλιση των γράφων καταχώρησης, αλλά ούτε αυτοί έχουν την αναλογή εντολή. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια εντολή και έχει γίνει μια αρχή. Κοιτώντα τι έχει γίνει στο 2010 με την Βελγική Προεδρία, ακούσαμε το επιχειρήμα ότι τα έγγραφα καταχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να έχουν καλύτερη ασφάλιση γιατί έτσι θα γλιτώσουμε πάρα πολλά προβλήματα και στην ομάδα εργασίας ε, του Συμβουλίου που ασχολείται με πλαστά εγγράφα, έγγραφα έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Υπάρχουν και κάποια έγγραφα εργασίας. Βλέποντας λοιπόν τι γίνεται εδώ θα πρέπει να υπάρξει παγκόσμια εναρμόνιση, να υπάρχουν δηλαδή Τέτοιε κατευθυντήριες γραμμέ ε, για όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα, αλλά προσπαθούμε να κοιτάξουμε αν μπορούμε να ορίσουμε και προδιαγραφέ και για τέτοια έγγραφα καταχώρηση έγγραφα πηγή. Στην Ευρώπη βλέπουμε ότι υπάρχει νομοθεσία για τα διαβατήρια, για τις θεωρήσεις, τα έγγραφα παραμονής και τώρα περιμένουμε λοιπόν ακόμα να υπάρξει κανονισμός σε ό,τι αφορά τα έγγραφα πήγη, τα έγγραφα καταχώρηση, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα διαβατήρια που κυκλοφορούν. Μία άλλη σημαντική ερώτηση την οποία θα έπρεπε να θέσουμε. Υπάρχουν πλέον εκτήματα για να γίνει εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ε, εγγράφων ε, καταχώρησης εγγράφων πήγης. Εμείς στο Project Fidelity θεωρούμε ότι ναι, υπάρχει προστιθέμενη αξία. Μία δεύτερη ερώτηση που θα έπρεπε να θέσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει και μία εναρμονισμένη διαδικασία έκδοση τέτοιων ε, εγγράφων πηγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί μόνο με την καλύτερη ασφάλιση των εγγράφων αυτών μπορούμε να κάνουμε καλύτερη, καλύτερους ελέγχους. Αν δεν υπάρχει ε, εναρμονισμένη διαδικασία έκδοσης, δεν θα σημειωθεί μεγάλη πρόεδρος. Και τέλος, ε, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων με κάθε σεβασμό φυσικά της ιδιωτικής σφαίρας σε ό,τι αφορά πληροφορίες για τέτοια έγγραφα καταχώρησης και τονίζω και πάλι το θέμα της ιδιωτικής σφαίρας το οποίο προστατεύεται. Παίζει σημαντικό ρόλο. Πραγματικά θα πρέπει να δεθούν κάποια ελάχιστα πρότυπα για τα έγγραφα αυτά προκειμένου να υπάρχει καλύτερη σύνδεση μεταξύ του εγγράφου ε, της πράξης γέννησης και του ατόμου που στη συνέχεια μετά από κάποια χρόνια ζητά ταξιδιτικό έγγραφο. προστατεύοντας παράλληλα την ταυτότητα του πολίτη. Η ταυτότητα και η υπηκότητα του πολίτη θα πρέπει πάντα να προστατεύεται και με την καλύτερη ασφάλιση των εγγράφων ε, καταχώρησης ε, θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Τέλος, να πούμε ε, ότι τα ηλεκτρονικά διαβατήρια λειτουργούν πιο εύκολα και πιο ομαλά και πιο γρήγορα και σε ό,τι αφορά την έκδοση εγγράφων καταχώρησης και την καλύτερη ευρωπαϊκή ρύθμιση θα έπρεπε να υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό ε, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε μόνο μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. So, όπως σας είπα, το πρόγραμμα Fidelity περιλαμβάνει έναν όμιλο 18 χωρών και ιδιωτικό και ε, δημόσιο τομέα, ε, εμπλέκονται αρχές, πανεπιστήμια κτλ. Τα πρώτα απορίσματα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Μέχρι το 2016 θα ε, συνεχιστεί το έργο αυτό και σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήσεις σε ό,τι αφορά τα έγγραφα καταχώρηση κτλ θα τα εξετάσει το πρόγραμμα Fidelity. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις και τώρα έχουμε χρόνο για συζήτηση. Έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Πριν να περάσουμε στο τρίτο μέρος της ακρόασης που θα ξεκινήσει στις 11 παρατέταρτο. Ο κύριο Κοέλιο, από ό,τι έχω καταλάβει, θα ήθελε το λόγο, εισηγητή, για να κάνει κάποιε ερωτήσει. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλες τις παρουσιάσεις, ήταν πολύ χρήσιμες. Στον ε, κύριο Τούντοράτς θέλω να πω ότι είμαστε πολύ καπνοποιημένοι που τελικά θα υλοποιηθεί το ΣΥΣ2, θα αρχίσει να λειτουργεί. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το πώς επιλέξατε αυτό το project και ασκήσατε την ε, ε, ηγεσία σας με ένα πολύ ρεαλιστικό τρόπο. Νομίζω ότι τα δύο πράγματα που άλλαξαν την ιστορία του δύο ήταν όταν εσείς αναλάβατε το έργο αυτό και όταν ε, δημιουργήθηκε και το Συμβουλίο Διαχείρισης και συμμετείχαν και τα κράτη-μέλη στο project. Επίσης, ε, καλωσορίζω τον κύριο Γκάρκοφ θα μεταβούμε στην υπηρεσία στα τέλη Απριλίου. Όπως ξέρετε, από το 2002 με την έκθεσή μου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε να δημιουργηθεί αυτή η υπηρεσία. Είμαστε ικανοποιημένοι λοιπόν. Πού ασχολείστε με το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν ε, θα απαντήσουν ε, ο κύριος Τούντερος ή ο κύριος Γκάρκοφ, αλλά έχω μια ερώτηση. Ο οργανισμός του προβλέπει μία εκστρατεία πληροφόρησης ε, προκειμένου το κοινό να ενημερωθεί σχετικά με τους ε, στόχους ε, των αποθηκευμένων δεδομένων ε, και των δικαιωμάτων ε, των πολιτών. Δεν ξέρω τώρα η Κομισιόν ή η Υπηρεσία είναι αρμόδια για το θέμα αυτό. Έχει γίνει κάτι σχετικά με αυτή την ενημέρωση, με αυτή την εξτρατή ενημέρωση, μπορείτε να με ενημερώσετε Κύριε Ρέχνερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση σχετικά με τη μελέτη. Εδώ και χρόνια εγώ έλεγα ότι το πρόβλημα είναι αυτό που δηλώσατε εσείς, το θέμα της καταχώρησης. Και επίσης τα πορίσματά σας συνάδουν όσα έχουμε ήδη πει στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και χαιρόμαστε που το συνειδητοποιούμε αυτό. Παρ' όλα αυτά είπατε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Τι θέλω να μου πείτε γιατί. Τι λείπει. Και πότε πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τις τελικές αξιολογήσεις της μελέτης αυτής. Και τέλος, κύριε Μπέλσερ. Σύμφωνα πολύ με όσα είπατε, το είπα και εγώ χτες. Στην έναρξη της ακρόασης, ο πιο αδύναμος κρίκος της ασφάλειας των διαβατηρίων είναι αυτά τα έγγραφα τα breeder documents. Το πρόβλημα είναι ότι είναι διαφορετικός ο πολιτισμός στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ε, κράτη-μέλη όπου υπάρχει υποχρέωση για δελτίο ταυτότητας, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη δεν υπάρχει. Υπάρχουν χώρες όπου τα αποτυπώματα μπορούν ε, να μπουν ε, στο δελτίο ταυτότητας, ενώ υπάρχουν άλλες χώρες που τα αποτυπώματα συνδέονται με το αν έχει κάποιος ποινικό μητρό. Συμφωνώ λοιπόν με όσα είπατε. Η ερώτηση μου είναι, τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί, ορθώ είπατε ότι ο ΙΚΑΟ δεν έχει εντολή για να ασχοληθεί με αυτό το θέμα των breeder documents στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιορίζεται από τις συνθήκες. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για το θέμα αυτό, είναι εθνικό ζήτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή, πέρα από το να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο, προκειμένου να ανταλλάξουμε πρακτικές και να θεσπίσουμε κατευθυντήριε γραμμέ. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που μα εξηγήσατε τόσο καλά. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σίπελ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο συγκεκριμένε ερωτήσει έχω να κάνω, αλλά θα ήθελα επί τη αρχή να κάνω μια προκαταρτική παρατήρηση. Δεν είμαι βέβαιη αν ξέρουμε τι κάνουμε, ότι ξέρουμε τι κάνουμε, αν μια μέρα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε δακτυλικά αποτυπώματα και βιομετρικά στοιχεία από όλους τους πολίτες μας, τουλάχιστον από τεχνικής άποψης, να είμαστε δηλαδή σε θέση τα στοιχεία αυτά να τα θέσουμε σε σύνδεση με άλλα στοιχεία για την δημιουργία προφίλ δεν αισθάνομαι και πολύ άνετα, να σας πω την αλήθεια. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καταρχάς προς τον κύριο Λέχνερ. Είπατε από πού προέρχονται τα, ε, τα φιλικά αποτυπώματα των παιδιών που πήρατε. Οι γονείς των παιδιών, θα ήθελα να ξέρω, είναι ενημερωμένοι ότι τα αθλητικά αποτυπώματα των παιδιών τους έχουν χρησιμοποιηθεί για, την, ε, για τους σκοπούς αυτούς, για τη μελέτη αυτή. Και προς τον κύριο Μπέλτζερ μιλήσατε για μια τάξη μεγέθους, για το πόσα άτομα ενδεχομένως ε, έχουν πραγματικό διαβατήριο, όμως, ε, το οποίο όμως έχει βασιστεί σε λανθασμένα πλαστά έγγραφα καταχώρησης. Τι άτομα είναι αυτά, ποια άτομα έχουν τέτοια διαβατήρια, είναι παράνομοι, ε, άτομα που διαμένουν απλά παράνομα στις χώρες αυτές. Πείτε μας λίγα λόγια. Eh Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχάρω όλους όσους, ε, όσοι έλαβαν το λόγο για την ποιότητα των παρεμβάσεών τους, για τη μετάβαση στο ΣΥΣ2. Την αναμέναμε βέβαια, είμαστε ικανοποιημένοι από όσα ακούσαμε, θα θέλαμε όμως να μας πείτε πώς συνδέεται τη φύλαξη των συνόρων με την εργασία σας. Ο κύριος Τοντεράς, τον οποίο συγχαίρω, τον ερωτώ το ζητώ να μας πει κάτι παραπάνω για τον νοτικό χάρτη για το πρόγραμμα που έχετε φέτος. Κύριε Λέχνερ, έχει, και να συγχαίρω και εσάς για την μελέτη που μας παρουσιάσετε. Έχετε την πρόθεση να τη δημοσιεύσετε για να υπάρχει επίσημα. Δεν θα έχετε βέβαια σήμερα τα γραπτά στοιχεία, αλλά η Κομισιόν σκοπεύει να τη διαδώσει, να τη γνωστοποιήσει και προς τον κύριο Μπέλζερ το πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε είναι φυσικά σημαντικό τα λεγόμενα breeder documents είναι φυσικά κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και η Ευρωπόλ θα μας τα πει όταν λάβει το λόγο αλλά όταν δίνετε αριθμούς για τη Γαλλία γιατί αναφερθήκατε στη Γαλλία πολλές φορές λέτε ότι υπάρχει ένα με 1,5 εκατομμύριο πλαστά διαβατήρια ε, επί συνόλου 6. Αυτό σημαίνει πάνω από 20% πλαστών διαβατηρίων στη Γαλλία. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Πού βασίζεστε. Έχω και εγώ αριθμούς. Και έγινε λόγος για αυτό το θέμα στην Ολομέλεια. Εγώ έχω άλλους αριθμούς. 20% είναι τεράστιος αριθμός. Για το 11 έχω στοιχεία από τη Γενική Διεύθυνση της Αστυνομίας των Συνόρων και λέει 233 επίσημα στοιχεία είναι αυτά, όχι άρθρο από τον τύπο, 233 πλαστά, 60 για διάφορες απάτες εκτός από ολόκληρα διαβατήρια είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό γενικότερα από 20% γιατί εμείς έχουμε στη Γαλλία έναν υπεύθυνο για κάθε αστυνομική διεύθυνση για τις απάτες και τα πλαστά, τις πλαστογραφίες. Δεν πρέπει λοιπόν να βασιζόμαστε σε ένα άρθρο στον τύπο που έχει ψεύτικα στοιχεία. Δεν αρνούμε ότι υπάρχουν πλαστογραφίες στη Γαλλία, αλλά οι αριθμοί που μας δίνεται είναι τελείως λανθασμένοι. Thank Uh, Ευχαριστώ. Προσπαθώ να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Και νομίζω ότι έχω κάποιες ερωτήσεις για το συς Σε ποιον ανήκει ο κώδικας και ποιος μπορεί να το διαχειριστεί. Ποιος μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή, αν τελικά προσταξουμε σε εξωτερική βοήθεια, θα πρέπει να πληρώσουμε, σε εξωτερική ανάθεση, να πληρώσουμε πάρα πολλά χρήματα στο μέλλον. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα επίπεδα, μπορούμε να έχουμε νέε διαπαφέ στον κώδικα. Με προγράμματα που δεν έχετε ακόμη σκεφτεί μέχρι σήμερα, για το μέλλον δηλαδή. Αν δεν μπορεί να ανοίξει ο κώδικα σε διαφορετικά επίπεδα, θα αναγκαστείτε να αγοράσετε ένα τελείω καινούριο πρόγραμμα και αυτό θα κοστίσει πολύ περισσότερα από όσο μπορούμε να διαθέσουμε. Και ποια είναι η πλατφόρμα του προγράμματος. Αυτές ε, τις ερωτήσεις έχω. Ευχαριστώ. you, Ευχαριστώ κύριε Γκιόν. Για να καθεσυγάσω την κυρία Ματιέ. Αν ε, υπάρχει καταπολέμηση αυτών των ψεύτικων ε, εγγράφων, των printed documents στα κράτη-μέλη στο παρελθόν, νομίζω ότι θα υπάρχει και στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί αναρωτιόμαστε και θέτουμε... Μάλλον ε, βλέπουμε τις διάφορες τεχνολογικές πτυχές που αφορούν τα θέματα της μετάπτωσης, Και είναι ενδιαφέρον ε, να ακούμε, παραδείγματο χάρη, το ότι αν ε, ένα παιδί είχε λερωμένα χέρια, αυτό θα μπορούσε να έχει επίπτωση στην ποιότητα των δακτυλικών του αποτυπωμάτων. Δηλαδή, αφενός να συζητούμε αυτό και από το άλλο να συζητούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα θέμα σχετικά με τα δεδομένα για κινδύνους ε, που ενέχονται. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια τεράστια γκάμα γάμα θεμάτων. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, για αυτό το θέμα των αποτυπωμάτων θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις, γιατί νομίζω ότι όλους μας εντυπωσίασε αυτό που μας είπατε για την ηλικία των παιδιών, τη στιγμή που πρέπει να πάρουμε τα αποτυπώματα και πώς ε, τελικά μπορούμε να καθορίσουμε με σαφήνεια αυτό ταυτότητα των παιδιών. Ε, πώς ε, έχει καθοριστεί το θέμα της ηλικία ε, και σε σχέση με άλλους φακέλους. Το αν είναι κάποιος ενήλικος ή όχι έχει να κάνει με το αν καθορίζουμε την ηλικία. Sí, Mr. Bronx. Yes, as a child I was wonderful. Όταν ήμουν μικρός δεν καταλάβαινα γιατί έπρεπε να πλένω τα χέρια μου και τώρα ξέρω για να μου παίρνουν τα αποτυπώματα. Το ΣΥΣ 2 θα χειρίζεται λέει 100 εκατομμύρια δελτία σε σύγκριση με μόνο 60 προηγουμένως. Γιατί χρειάζονται τόσο πολύ περισσότερα δελτία και νου στοιχεία περιλαμβάνει, με τι κριτήρια συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία κάποιου. Όλα τα δελτία είναι από ανθρώπους εκτός ένωσης που έχουν ζητήσει να μπουν σε αυτήν ή που έχουν μπει. Ε, Μήπω αποκλείονται ορισμένες χώρες μέλη. Είναι άνθρωποι που έχουν ζητήσει θεώρηση, ορισμένοι που είναι ύποπτοι για οργανωμένο έγκλημα ή για τρομοκρατία ή πολιτικώ αντιφρονούντες. Και πώς χρησιμοποιούνται τα δελτία, σε ποιον δίνονται, χορηγούνται και σε τρίτες χώρες. Τώρα, ο κύριο Λέχνερ είπε, ελπίζω να το κατάλαβα καλά ή να το άκουσα σωστά, ένα εκατομμύριο κάτοικοι της Ολλανδίας έχουν πλαστά διαβατήρια και αναφέρατε και γαλλικά πλαστά διαβατήρια. Όχι, λάθος έκανα, λάθος έκανα, πάντων. Διορθώστε με. Και μεταξύ 500.000 και ενός εκατομμυρίου πλαστών εγγράφων, δεν ξέρω αν είναι έγγραφα πηγής Breeder Document στη Γαλλία. Φαντάζομαι ότι οι αριθμοί αυτοί ισχύουν περίπου πάνω κάτω και στις άλλες χώρες μέλη. Όχι σε όλες βέβαια γιατί δεν πηγαίνουν περισσότεροι μετανάστες στις φτωχότερες χώρες. Αυτά είναι μόνο όσα έχουν αποκαλυφθεί. Μπορεί να υπάρχουν με υψηλότεροι αριθμοί από ανθρώπους των οποίων δεν γνωρίζουμε τα στοιχεία. Και φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που χρησιμοποιούν πλαστά διαβατήρια είναι παράνομοι μετανάστες ή εγκληματίες που θέλουν να διαφύγουν από τη δικαιοσύνη. Πάλλον όμως περισσότεροι μετανάστες. Τέλος, να μου το επιβεβαιώσετε, τέλος, ποιος θεωρείται υπεύθυνο για την πλαστογραφία. Μιλάμε για πολύ μεγάλης κλίμακας οργανωμένο έγκλημα ή γίνονται τα πράγματα σε μικρή κλίμακα και τοπικά. Γιατί η πλαστογράφηση θα μπορούσε να λύσει το συλλογικότερο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ωραία, έγινε ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων, Μερικά ήταν πολύ, μερικές ήταν πολύ συγκεκριμένες και θα απαντήσουν οι πανελίστε με τη σειρά, με την ίδια σειρά με την οποία έλαβαν το λόγο. Πρώτος ο κύριος Τουντεράτς λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και όλα τα άτομα που πήραν το λόγο και έθεσαν πολύ καλές ερωτήσεις για να απαντήσω τις ερωτήσεις με τη σειρά για το ΣΥΣ 2. Καταρχάς να απαντήσω στον κύριο Κοέλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πάρα πολύ γενικά σας λόγια. Να σας πω για την εκστρατεία ενημέρωση Όντως ε, προβλέπετε τέτοια εκστρατεία και πριν από κάποιους μήνες ε, αναπτύξαμε τη σχετική εκστρατεία ενημέρωση. Μέχρι σήμερα Έχουμε φυλάδια, παραγωγή, πόστερ ε, και ένα μικρό βιντεάκι. Πρόκειται για ένα κοινό project με τα κρατημέλη. Άρα η όλη ιδέα είναι ότι τώρα βρισκόμαστε σε φάση εμ, παροχής του υλικού που έχει παραχθεί και μαζί με τα κρατημέλη και τους αρμοδίους διανέμουμε το υλικό αυτό, γιατί τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την ε, παροχή του υλικού αυτού στην επικράτειά τους. Οι πολίτες μας πρέπει να γνωρίζουν το συς και όλοι οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για το τι κάνει πλέον το συς Από πλευράς μας προτιμάζουμε τέτοια διανομή του υλικού των πληροφοριών αυτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σίγουρα θα περιληφθεί στο δίκτυο αυτό. Μόλις λοιπόν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή σε μια-δύο θα αποστείλουμε το υλικό αυτό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από πλευρά περιεχομένου δίδεται μια σωστή αποτύπωση των δικλείδων ασφαλείας, των μηχανισμών που έχουν οι πολίτες για τη διόρθωση των στοιχείων τους ενδεχομένως. Τώρα, τέθηκε ένα ερώτημα, νομίζω, για την ε, μετανάστευση του συστήματος, το ρόλο των ε, συνοριοφυλάκων, οι οποίοι σίγουρα χρησιμοποιούν και αυτό το σύστημα, περιλαμβάνονται στο σύστημα, όπως και άλλες αρχές εφαρμογής του νόμου. Είπαμε ότι στις 9 Απριλίου και στις 9 Μαΐου θα είναι οι ημερομηνίε για, για την ολοκλήρωση τη περίοδου ε, επιτήρηση και από εκείνη την ημερομηνία και μετά θα ισχύει το ΣΥΣ 2, πάει το ΣΥΣ 1. Και ύστερα ελπίζουμε να λειτουργήσει απρόσκοπτα, χωρί προβλήματα. Δεν υπάρχει άλλο σημείο ελέγχου το οποίο προβλέπεται μετά τις 9 Μαΐου. Άλλο ένα στοιχείο σε ό,τι αφορά την σαφή εξέλιξη ε, ή τα στοιχεία τα οποία προστίθενται είναι τα βιομετρικά στοιχεία. Αυτό βάσει της έκθεσης που θα υποβάλει καταρχάς η Επιτροπή στο Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο, συγγνώμη. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των βιομετρικών στοιχείων. Ένα άλλο θέμα που ερωτήθηκε ήταν το θέμα της ιδιοκτησίας του κώδικα. Η Επιτροπή είναι ιδιοκτήτης του κώδικα ως τώρα ήταν υπεύθυνη για το ΣΥΣ1 και ως ε, αναθέτουσα αρχή για το ΣΥΣ2. Είμαστε οι ιδιοκτήτες και φυσικά θα το διαβιβάσουμε. Μπορούν να γίνουν τροποποίησεις βεβαίως αν είναι συμφωνηθούν κάποιες εξελίξεις από τους τελικούς χρήστες. χρήστες η του συστήματος είναι δυνατές. Ποια είναι η πλατφόρμα του ΣΥΣ2. Πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο έχει κατασκευαστεί, έχει παρασκευαστεί. Δεν είναι κάτι το οποίο διτίθεται ευρέω. Αύξηση των ε, δυνατοτήτων. Γιατί? Όντω, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ένα από τους βασικούς παράγοντες για την αύξηση των καταχωρήσεων. Όχι μόνο αύξηση σε αριθμό, αλλά και η χρήση του συστήματος, ξέρετε, καθορίζει το μέγεθος. Εκατό εκατομμύριο, γιατί το 2010 έγινε μία μελέτη η οποία εξέτασε τις τάσεις τις εξελεκτικές σε ό,τι αφορά την αύξηση καταχωρήσεων ένα κράτος μέλος και αποφασίσαμε ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα υπήρχε αύξηση κατά 75 εκατομμύρια. Άρα εμείς είχαμε προβλέψει αύξηση κατά 100 εκατομμύρια. Θεωρούμε λοιπόν ότι το σύστημα είναι αρκετά μεγάλο για να μην χρειαστεί στο εγγύς μέλλον άλλη αύξηση του δυναμικού, άλλη αύξηση των ικανοτήτων και να μπορεί να παρέχει ένα σταθερό περιβάλλον για τους χρήστες, κριτήρια για το ποιοι περιλαμβάνονται στο σύστημα και ευρωπαϊκή, ε, υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Τα αντικείμενα είναι πολύ διαφορετικά σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, πλοία, πιστοτικές κάρτες κλεμμένες, κλεμμένα ταξιδιωτικά έγγραφα, Υπάρχουν πάρα πολλοί ειδών καταχωρήσεις λοιπόν στο σύστημα σε ό,τι αφορά τα άτομα, ναι, υπήκοοι τρίτων χωρών που μπαίνουν στο χώρο Σέγγεν, αλλά και Ευρωπαίοι υπήκοοι σε περίπτωση που έχουν ε, εκδοθεί κατά αυτόν ε, εντάλματα σύλληψης αλλά και άτομα τα οποία αγνοούνται, παιδιά τα οποία αγνοούνται για παράδειγμα. Άρα έχουμε και αυτό το πλέον έκτημα σε ό,τι αφορά αγνοούμενα άτομα. Αυτή νομίζω ήταν η τελευταία ερώτηση. Α, μάλιστα. Κατά πόσον οι πληροφορίες ε, του συς μπορεί να μεταφερθούν σε άλλες χώρες. Όχι. Αυτό ορίζεται με ασφαλιστική δικλίδα στην νομοθεσία. Για τη δημοσίευση τώρα της ε, μελέτης, νομίζω το ρώτησε ο κύριος Λέιχνερ. Και πάλι πρόκειται για ένα, μια σύμβαση της Γενικής Διεύθυνσης Home. Εμείς ζητήσαμε να γίνει η μελέτη αυτή και σας διαβεβαιώ ότι όταν λάβουμε την τελική έκθεση θα τη μοιραστούμε και με το DPS και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, θα παρακαλούσα και τους υπόλοιπους ομιλητές να είναι σύντομοι. Ο κύριος Γκάρκοβ για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σίγουρος ότι αφήθηκε κάτι αναπάντητο. Όμως, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις σχετικά με το ΣΥΣ, μπορώ να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο κύριος Τουντοράτς. Δηλαδή ότι στο τέλη Μαΐου ολοκληρώνεται η περίοδος παρακολούθησης του συστήματος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθέσει όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση του συστήματος, την υπηρεσία που θα έχει πρόσβαση σε αυτά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το θέμα των εξέλιξεων και τις αλλαγές ε, στα συστήματα. Ανάλογα και με τις ανάγκες των κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριε Ζλέκνερ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και εγώ να απαντήσω στις ερωτήσεις μία-μία. Καταρχήν για τη μελέτη όπου λέμε προκαταρκτικά πορίσματα σήμερα, τι λείπει. Αυτό που λείπει είναι η ίδια η μελέτη, γιατί κάναμε τους ελέγχους και τις μετρήσεις ε, και είδαμε πόσο καλά λειτουργούν όλα αυτά, όμως όλα αυτά πρέπει να τεκμηριωθούν. Και είμαστε ικανοποιημένοι που βρήκαμε εδώ την ευκαιρία για να παρουσιάσουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι αρκετά αξιόπιστα, όμως η ίδια η μελέτη λείπει. Πρέπει να γίνει λοιπόν αυτό. Τώρα το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι θα έχουμε την τελική μελέτη τον Αύγουστο. Και υπήρξε και μια ερώτηση, γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό σχετίζεται με τον ευαίσθητο χαρακτήρα των ε, αποτυπωμάτων και με άλλα ζητήματα εν μέρη υπήρξε εις βάθος μελέτη για το πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων που υπάρχουν στην Πορτογαλία, υπό ποιες συνθήκες και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Και νομικά πρέπει να το ρυθμίσουμε αυτό. Ε, συμμετείχε και ο επόπτης ε, προστασίας των δεδομένων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πορτογαλίας και η κυβέρνηση της Πορτογαλίας που συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα, αλλά έπρεπε και η Πορτογαλική κυβέρνηση να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα για το πώς ε, θα περιορίσει το χώρο που μπορούσε να η μελέτη και κατόπιν εν μέσω οικονομικής κρίσης η πορτογαλική κυβέρνηση επανεκλέχθηκε έπρεπε λοιπόν να ξαναρχίσει μια διαδικασία από την αρχή με νέα κυβέρνηση. Αυτό καθυστέρησε την όλη διαδικασία πάρα πολύ και τελικά χαιρόμαστε που δεχτήκαμε την έγκριση και περιμένουμε τον Αύγουστο να έχουμε τα αποτελέσματα σε έγγραφο. Επόμενη ερώτηση. Έχει νόημα να παίρνουμε αποτυπώματα παιδιών όλων των ηλικιών. Θα απαντήσω στα αγγλικά. Δεν το ερευνήσαμε αυτό το θέμα στην μελέτη. Τεχνικά μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να γνωστούν αποτυπώματα και από πολύ μικρές ηλικίε. Οι Πορτογάλοι εξαντλητικά παίρνουν ε, αποτυπώματα των πολιτών τους από πολύ μικρές ηλικίε ήδη. Τώρα για τον αν έχει νόημα δεν νομίζω ότι θα αποφασίσουμε εμείς εδώ. Απλώς ε, ρίχνουμε κάποιο φως στις τεχνικές, ε, τεχνολογικές ε, δυνατότητες και λέμε ότι μπορούν να γνωριστούν τα αποτυπώματα ακόμη και ανθρώπων μικρής ηλικία. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τώρα το θέμα της της ηλικία ή όχι. Ερώτηση. Αν είχαν ενημερωθεί οι γονείς των παιδιών για τη χρήση των δεδομένων ελέγχθηκε αυτό και πρέπει να ελεγχθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασία των δεδομένων, δηλαδή τις πορτογαλικές αρχές που έχουν το σύνολο των δεδομένων στην κατοχή τους. Και φυσικά γι' αυτό χρειαστήκαμε για τόσο πολύ χρόνο να έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες. Ο περιορισμένο καθήκον της μελέτης ε, του GRC σε μόνο ηλεκτρονικά τυπώματα που δεν ε, μπορούν να σχετιστούν με τα άτομα και δεν μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε όλη τη βάση δεδομένων, αλλά μόνο σε ένα δείγμα της βάση δεδομένων. Υπήρχαν περιορισμοί λοιπόν σε αυτό και θα ήθελα να παραμείψω και πάλι στις πορτογαλικές αρχές και δεν μπορώ να μαντέψω τώρα αν ενημερώθηκαν ή όχι οι γονείς των παιδιών. Τουλάχιστον οι αρχές όλες είχαν ενημερωθεί και είχαν συνενέσει Νομικά ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα. Ανατέθηκε αυτή η μελέτη στο JRC μόνο από συγκεκριμένε συνθήκες. Οι άλλε ερωτήσει για τη δημοσίευση έχουν απαντήθει. Υπήρξε και μία ερώτηση για το αν θα χρησιμοποιηθούν τα αποτυπώματα για να βρεθεί αν κάποιος ε, έχει κλείσει τα 18 ή όχι. Ούτε αυτό είναι το αντικείμενο της μελέτης δεν μπορούμε να πούμε τίποτα σχετικά με τη δυνατότητα να ανεχρεύσουμε την ηλικία από το αποτύπωμα. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα. Ίσως ε, χρειάζεται να αποσαφινιστεί συζήτηση στο μέλλον, όμως εγώ δεν μπορώ να πω ότι το αποτύπωμα αυτό σε ένα παιδί 14, 15, 16 χρονών. Δεν ε, μπορούσαν να δουν πόσο θα μεγαλώσουν τα παιδιά μέχρι να φτάσουν στο 18. Πρόεδρος, ευχαριστώ. να ακούσουμε και τον κύριο Μπέλσερ, τον τέταρτο προστίκλημένο μας. Αλλά πριν από αυτό, μήπως να δούμε αν υπάρχει κάποια πρόσθετη ερώτηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις με τη σειρά που τέθησαν. Ε, όντως, κυρία, ξεκινήσαμε με ένα άρθρο στην Παριζιέν του 2011 όπου αναφέρθηκαν τα θέματα αυτά και το ζήτημα για το πόσα ηλεκτρονικά διαβατήρια έχουν εκδοθεί βάσει εσφαλμένων πλαστών εγγράφων πηγή. Συζητήθηκε τον Απρίλιο του 2012 στο Κοινοβούλιο. Το γεγονός και το ερώτημα το κατά πόσον ισχύουν τα αριθμητικά στοιχεία έχει τεθεί και στους υπαλλήλους που ασχολούνται με τέτοια θέματα πλαστών διαβατηρίων και μας είπαν ότι είναι σημαντικός αριθμός διαβατηρίων. Τώρα κατά πόσο είναι 4.000, 6.000, 8.000 τα διαβατηρία δεν το ξέρουμε. Και επίσης ε, κάναμε σχετικές ερεύνες στην Ολλανδία σε μια σύντομη χρονική περίοδο περίπου 1.000 άτομα με παρουσιάστηκαν με γαλλικά ε, αυθεντικά διαβατήρια στη Χάγη και κατά την καταχώρηση στα, στις Αρχές πρέπει να δώσει κανείς και ένα, μια πράξη γέννησης και εκεί προέκυψε ότι ήταν πλαστά τα έγγραφα της πράξης γέννησης. Και οι αρχές αυτό μπορούσαν να το διαπιστώσουν με ένα μικρό ε, μεγεθυντικό φακό του ενός ευρώ. Άρα οι Ολλανδικές αρχές ανέφεραν ότι περίπου χίλια άτομα διαμένουν στις κάτω χώρες, τα οποία έχουν ε, ε, προέλευση από την Βόρεια Αφρική, από την Καραϊδική και έχουν διαμείνει επί σειρά ετών στην Γαλλία παράνομα και μετά με αυτή την ε, εύκολη παραχάραξη είδαν την ευκαιρία τους προκειμένου να εκδώσουν ένα αυθεντικό διαβατήριο βάσει όμως πλαστού εγγράφου καταχώρησης. Και από τις χίλιες περιπτώσεις ε, που διαπιστώσαμε στην Ολλανδία, 400 αντιδράσεις έχουμε και απαντήσεις έχουμε λάψει από τις γαλλικές αρχές, οι οποίες ε, επιβεβαιώνουν ότι όντως εκδόθηκε διαβατήριο βάσει πλαστών εγγράφων καταχώρησης και οι γαλλικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν για να ελαχιστοποιήσουν το πρόβλημα αυτό στο βαθμό του δυνατού ασφαλώς. Ε, ερώτηση εκτός μικροφώνου. 400 διαβατήρια όμως δεν είναι 1,5 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτό ε, το διαπιστώσαμε στο, στην Ολλανδία, 400 διαβατήρια. Και ακόμα και οι γαλλικές αρχές ε, ε, μίλησαν για άρθρα στις εφημερίδες που αναφέρουν μισό έως ένα εκατομμύριο τέτοια διαβατήρια. Τώρα, ε, είτε είναι 800.000, 600.000, 1 εκατομμύριο. Αυτός ο αριθμός ερευνάται από τις γαλλικές αρχές, αλλά είναι πάρα πολλά τα ηλεκτρονικά διαβατήρια γαλλικής ε, έκδοσης που έχουν εκδοθεί βάσει πλαστών ε, γράφων καταχώρησης. Κοιτάξτε, είναι ένα γνωστό παράδειγμα το, το, η περίπτωση της Γαλλίας, αλλά δεν συμβαίνει αυτό μόνο στη Γαλλία. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται αυτές οι παραχαράξεις ε, από άτομα τα οποία δεν έχουν δικαίωμα έκδοσης νόμιμου διαβατηρίου τέτοιου. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος και τώρα μπορούμε να κλείσουμε το τμήμα Τελειώνει και αυτό το μέρος στις 10 και 45 θα αρχίσουμε τον τρίτο θέμα με τον κύριο Νίλσεν, Γιάντεμπος και Μπουταρέλη αν παραμείνουν ανοιχτά ερωτήματα να τα δείξουμε τώρα. Αν όχι, διάλειμμα 10 λεπτά 1 τέταρτο και θα συνεχίσουμε στις παρατέταρτο.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 Υπότιτλοι last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 Γεια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

Magdalena

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την ε, τρίτη και τελευταία συζήτησή μας για τις περαιτέρω εξελίξεις. Και θα ακούσουμε τρεις προσκεκλημένους, ο οποίους θέλω να καλωσορίσω, τον κύριο Ζήλια Ζαντεμπούρ από το Κέντρο Μελετών για τις Σειράξεις τον κύριο Χέριν Κλίνσεν από τη Γαμμαδάλη Τεστορικών Υποθέσεων και τον κύριο Τζοβάνι Μπουταρέλη από το Γραφείο του Ευρωπαίου Πόπτη Προστασία των Δεδομένων. Και θα υπάρξουν και αντιδράσεις από την κυρία Ρενάτε Ζόμερ και τον κύριο Ιον Έντσου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ για την προσέλευσή σας εδώ και να δώσω τον λόγο στον κύριο Ζαντεμπό. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Θα σας παρουσιάσω τα κύρια ερωτήματα και τα πορίσματα μια μελέτης ε, που έχει να κάνει με τη βάση δεδομένων για φύση σύνορα και ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εκ μέρους της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ. Θα σας παρουσιάσω τα κυρία θέματα που εξετάζει αυτή η μελέτη, τα κυρία πορίσματα σχετικά με το πώς τα εφή σύνορα μπαίνουν στο σημερινό τοπίο των βασών δεδομένων. Ε, για τις ιστορικές υποθέσεις επίσης θα αξιολογήσουμε την πρωτοβουλία των φιών σύνορων και τις προκλήσεις ε, αυτής της πρωτοβουλίας για να ξεκινήσουμε με τα κυρία ζητήματα. Καταρχήν η μελέτη εντοπίζει τρία κυρία θέματα. Καταρχήν ε, το θέμα της αντιστρεψιμότητας, της αναγκαιότητας και, της, ε, ε, και του αυθεντικού χαρακτήρα. Ορισμένες από τις ε, προτάσεις που έχουν τώρα κατατεθεί έχουν ε, κυκλοφορήσει εδώ και καιρό. Αν σκεφτείτε το θέμα, το σύστημα εισόδου-εξόδου συζητήθηκε το 2004 από την Κομισιόν. Ε, το θέμα λοιπόν της, της αφορά τη δυνατότητα, οι εφαρμογές που έχουν εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξουν πορεία αν υπάρχουν νέες εξελίξεις. η αναγκαιότητα προκύπτει από το πρώτο, οι σημερινέ προτάσει για τι νέε βάσει δεδομένων συμπεριλαμβανομένων και των ευφυών συνόρων παρουσιάζονται ω απαραίτητε για να συμπληρώσουν παλιά μέτρα και έρχονται εδώ σήμερα για να συμπληρώσουν το ΣΥΣ και το ΒΙΣ αλλά αυτή η αναγκαιότητα σχετίζεται με τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών και με την καλή λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών μας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θέτει μελέτη. Τώρα, ο αυθεντικός χαρακτήρας ρωτά τα μέτρα που ε, προτείνονται, αντικατοπτρίζουν τις ε, νομικές υποχρεώσεις και τις αρχές και τις αξίες ε, που εγγράφονται στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Οι σημερινές προτάσεις και το πακέτο των ευφυών συνόρων ή κάποια άλλα συστήματα βασίζονται σε πρωτοβουλίες που έχουν θεωρηθεί από τέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Αυστραλία ή η ΕΠΑ. Τώρα το θέμα είναι ε, προσαρμόζονται στις δεμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά και ε, τους πολίτες και τους πολίτες των τρίτων χωρών σε ό,τι αφορά ορισμένα από αυτά τα θέματα, η μελέτη βασικά ρωτά ποιος ε, είναι ο προβλεπόμενος αντίτυπος των βάσεων ε, δεδομένων ε, και επιχειρηματολογεί ότι η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτικότητα είναι απαραίτητα θέματα που πρέπει να τεθούν, αλλά δεν αρκούν. Και μία από τις κύριες προτάσεις της μελέτης είναι ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα της εισαγωγής διακρίσεων και να υπάρξει δέσμευση για τη μη διάκριση σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ελέγχου συνόρων. Καταρχήν θα σας αναφέρω τα κύρια πορίσματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που τα, η πρωτοβουλία των ευφυών συνορών ε, εντάσσεται στο τοπίο των βάσεων δεδομένων. Υποθέτουμε ότι τα ευφυή σύνορα δεν μπορούν να εξεταστούν με μονομένα από τις άλλες πολιτικές. Ανήκουν στο συγκεκριμένο τομέα ιστορικών υποθέσεων, δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων, αλλά θα πρέπει να τα σκεφτούμε σε σχέση με τις ευρύτερες τάσεις. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε αυτή την έννοια του είναι επειδή έχει υπάρξει μία τάση να παρουσιάζεται κάθε νέο μέτρο που σχετίζεται με την επεξεργασία των δεδομένων για ε, λόγους δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων για να συμπληρωθούν ε, τα κενά ε, όμως παρουσιάζουμε και ποιες υπηρεσίες έχουν πρόσβαση σε αυτά. Ε, τώρα λοιπόν αναπτύσσουμε ένα τοπίο μέτρων που ε, μπορούν να υπερβαίνουν τα σύνορα και τις δικαιοδοσίες. Είχαμε και μία αξιολόγηση το 2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25 υφιστάμενων και μελλοντικών βάσεων δεδομένων όμως, ενώ μερικές φορές ε, αναφερόμαστε σε αυτές τις βάσεις δεδομένων ενό βάσεις δεδομένων δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων, δεν υπάρχει επίσημος ορισμός για το πώς θα πρέπει να είναι με τέτοια βάση δεδομένων. Και παρόλα αυτά η μελέτη υπογραμμίζει ότι υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία που μας επιτρέπουν να καταλάβουμε τις γενικές τάσεις πολιτικής. Αυτά τα κοινά στοιχεία είναι τα εξή. Καταρχήν, σχετίζονται με την ανταλλαγή δεδομένων ε, by default, εκ προγραμματισμού, εξορισμού. Ε, αυτό υποστηρίζεται από την αρχή της διαθεσιμότητας ε, και από την αρχή της διαλειτουργικότητας που ρυθμίζει τις πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ των συστημάτων. Όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι ούτε η διαλειτουργικότητα ούτε η διαθεσιμότητα είναι νομικές αρχές. Δεύτερον, έχουμε η εξέλιξη αυτών των βάσεων δεδομένων έχει να κάνει με την ε, επεξεργασία, την ευρία επεξεργασία των δεδομένων, την ευρία επεξεργασία των δεδομένων. Υπάρχουν ε, διαφορετικές βάσεις δεδομένων κατακαιρματισμένες και έτσι λοιπόν ε, είναι δύσκολο να προσφέρουμε την κατάλληλη προστασία των δεδομένων. Αυτό το αποκεντρωμένο ε, σύστημα μας παραπλανεί. Ε, αν ε, λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν επικαλυπτόμενες δυνατότητες τη συλλογή της ανταλλαγής και της πρόσβασης των δεδομένων, η έννοια αυτής της ευρείας διανομημένης επεξεργασίας των δεδομένων είναι μου ζήτησαν οι διερμηνείς να μιλάτε πιο αργά. Καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή είναι των δεδομένων, όπως έλεγα, είναι πολύ πιο ακριβής. Και φυσικά ε, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει τεχνικό όριο στην επεξεργασία των δεδομένων. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων. Ε, στον τομέα δικαιοσύνη και ιστορικών υποθέσεων. Ε, περισσότερα συστήματα επεξεργασία των δεδομένων στον τομέα ΔΕΗ έχουν πολλαπλού σκοπού. Δηλαδή, σχετίζονται με ένα τομέα πολιτική, αλλά δεν είναι αποκλειστικό αυτό ο σύνδεσμο, είναι προτιμητέο. Και αυτό ισχύει για την πρόσβαση στο ΒΙΣ από τι διοκτικέ αρχέ και γι' αυτό συζητάμε να ανοίξουμε την πρόσβαση των ε, διοκτικών αρχών στο σύστημα εισόδου-εξόδου. Επίση, βρίσκουμε σύνδεση σε σχέση μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ επιχειρησιακών και προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα χωρίζονται σε δύο μέρη. Καταρχήν έχουμε τα επιχειρησιακά δεδομένα και τα προσωπικά δεδομένα. Όμως αυτή η διάκριση έχει να κάνει με την ικανότητα των αξιωματικών του διοκτικών αρχών να προσωποποιήσουν τα δεδομένα για να χρησιμοποιηθούν για επιχειρησιακούς σκοπούς και εδώ τίθεται ένα ερωτηματικό όταν μιλάμε για τις εγγυήσει για τα άτομα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Τώρα, Βάσει των πορισμάτων αυτών, η μελέτη εντοπίζει τρία κυρία ζητήματα. Καταρχήν, Έχουμε την ε, εν μέρη υποβολή εκθέσεων που αναφέρεται στην επεξεργασία των δεδομένων. Ορισμένες δεξιότητες αναφέρονται, όπως σε παρακολουθώς χάρη στο απόφαση Προύμ, στο σύστημα υπόφαση Προύμ ή στο Eurodac και στο ΣΥΣ, όπως παρακολουθώς χάρη. Για άλλα συστήματα, όπως η Σουηδική Πρωτοβουλία, δεν έχουμε τέτοια συστήματα. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τον τρόπο που αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν σχεδιαστεί. Συχνά σχετίζονται με συγκεκριμένα γεγονότα, με παρελθόντα μέτρα, όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ικανοποιητική ε, δεν είναι ικανοποιητικέ οι αποδείξει που έχουμε. Επίση, πολλέ φορέ μετακινούμαστε στη μαζική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και αυτή είναι μια επιλογή που άλλοι εταίροι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα η Αυστραλία, έχουν επιδιώξει, κυρίω μετά τι επιθέσει τη 11 Σεπτεμβρίου. Όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση στο στάδιο αυτό ε, θα έπρεπε να ακολουθήσει με τέτοια εξέλιξη. Εδώ σα ε, δείχνουμε μία απεικόνηση για το τι εννοούμε με τη μαζική επεξεργασία. Έχουμε συμπεριλάβει και την πρωτοβουλία PNR τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σχετίζεται με τέσσερι διασυνοριακού ελέγχου. και πρέπει να καταλάβουμε ότι τα ΕΦΗ e σύνορα δεν είναι ένα μεμονωμένο μέτρο. Πρέπει λοιπόν να δούμε πόσο έχει αυξηθεί η επεξεργασία των δεδομένων σε σχέση με τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί που εξετάζουμε στα πλαίσια τη πολιτική ΔΕΗ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με την αξιολόγηση της πρωτοβουλίας των ευφύων συνόρων. Βασίζεται στην ανακοίνωση της ε, Κομισιόν. Ε, δεν θα αναφέρω τις τεχνικές πτυχές, νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει αργότερα. Πολύ σύντομα η πρωτοβουλία των ευφυών συνόρων να έχει τρει κύριε αλλαγέ ε, Καταρχήν την αυτοματοποίηση των συνεργειακών ελέγχων. Τα συμπολογιστικά συστήματα καλούνται να αντικαταστήσουν μια σειρά δράσεων στον έλεγχο των ταξιδιωτών. Δεύτερον, διεύρυνση τη εξεργασία των δεδομένων σε μια κατηγορία ταξιδιωτών που δεν είχαν ε, τεθεί στο στόχο στο το μέτρο, χάρη σε ταξιδιώτε που δεν χρειάζονται θεώρηση και επίση αντικοποίηση του ελέγχου για ταξιδιώτε όπου απαιτείται θεώρηση ανταλλαγή θεώρηση. Αυτά τα τρία απορρίμματα οδηγούν στο να συζητήσουμε τρία ζητήματα. Καταρχήν, ε, το να βασιζόμαστε σε αποδείξεις ε, που να καθορίζουν την αναγκαιότητα και επάρκεια των συστημάτων. Η πρωτοβουλία των εξύπνων συνόρων βασίζεται στα μέτρα που εν μέρει έχουν εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη όπως και στις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, κυρίω μέσω του προγράμματος θεωρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην περίπτωση του προγράμματος αυτού, Έχουμε σημαντική κριτική από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ότι κοστίζει πάρα πολύ το σύστημα, δεν είναι ε, καλά τα αποτελέσματα και το ερώτημα είναι πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αποτιμήσει αυτή τη μερική αποτυχία του όσων προσπαθούν να κάνουν οι νομές Πολιτείες και είναι ρεαλιστικό και επιθυμητό να εφαρμόσουμε τα μέτρα που προβλέπονται στην ε, πρωτοβουλία εφιών συνόρων μέσα στα χρονικά όρια που έχουμε θέσει. Δεύτερον, το κόστος των προτάσεων. Δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς, υπάρχει στη μελέτη, όμως διακυμαίνεται η εκτίμηση του κόστους το 8 η πρόταση της ανακοίνωσης της Κομισιόν προέβλεπε ε, για ένα κόστος 20 εκατομμύριων ευρώ για να συσταθεί ε, το σύστημα 6 ε, εκατομμύρια ετησίως για τη συντήρηση και φτάναμε λοιπόν στα 400 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Έτσι λοιπόν πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό του κόστους ε, για το σύστημα εισόδου-εξόδου και για το σύστημα εγγεγραμμένων ταξιδιωτών. Τώρα, επέκταση του ελέγχου για τους ε, αλλοδαπούς ταξιδιώτες. Εδώ λαμβάνουμε υπόψη ότι ελέγχονται οι ταξιδιώτες πριν, κατά τη διάρκεια μετά του, ταξιδιού, του, του ταξιδιού τους αυτό έχει σημαντικές προκλήσεις ε, που τίθεται από την πρωτοβουλία έξυπνων συνόρων. Αυτές οι προκλήσεις, όπως είπα προηγμένως, συζητούνται σε σχέση με δύο θέματα. Καταρχήν, η προστασία των δεδομένων ε, και το απόρριτο και το θέμα της εισαγωγής διακρίσεων. Η προστασία των δεδομένων είναι απαραίτητα, αλλά δεν αρκεί. Φυσικά, η επεξεργασία των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα ε, πρέπει να τη δούμε με το θέμα του απόρριτου που ε, φτάνει στο να δείξει την ιδιωτική ζωή, όπως ε, λέει το άρθρο 7 τη Σύμβαση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης σχετίζεται με την αρχή της ασφάλειας δικαίου που έχει να κάνει με την δυνατότητα προσφυγής και επίσης οι διάφορα συστήματα επεξεργασία των δεδομένων θέτουν ερωτήματα σε σχέση με την αναγκαιότητα και τα κριτήρια του περιορισμού του σκοπού. Το δεύτερο τμήμα των προκλήσεων έχουν να κάνουν με το θέμα της μη εισαγωγή διακρίσεων. Φυσικά, οι υπηκοί τρίτων χωρών δεν καλύπτονται επί της αρχή από την προστασία που προσφέρει η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μη εισαγωγή διακρίσεων βάση εθνικότητα, όμω υπάρχουν κάποιε διατάξει που ισχύουν για του υπηκόους τρίτων χωρών όταν μιλάμε για την εισαγωγή διακρίσεων στο συνοριακό κώδικα Σέγγεν. Η εθνικότητα και το νομικό καθεστώ δεν μπορεί να θεωρηθούν ε, ω ε, παράγοντε, αλλά οι υπήκοοι τρίτων χωρών προστατεύονται από την εισαγωγή διακρίσεων για θέματα όπω είναι η ηλικία, ο γενετήσιο προσανατολισμό, η θρησκεία, οι πολιτικέ απόψει κτλ. Όμως πρέπει να δούμε πόσο δύσκολο είναι να διακρίνουμε την εισαγωγή διακρίσεων βάσει της εθνικότητας ή ε, βάσει της φυλής. Επίσης, ε, το βασικό, η βασική λογική για το διασυνοριακό έλεγχο γίνεται βάσει της εθνικότητας ε, και ε, η εθνικότητα δεν θα πρέπει να αποτελέσει έναν τρόπο εισόδου εισαγωγής διακρίσεων άλλης μορφής. Και το βασικό θέμα εδώ είναι η αυτοματοποίηση ε, των ε, συνοριακών ελέγχων. Η μελέτη τονίζει ότι το θέμα ε, της δημιουργίας προφίλ πρέπει να εξεταστεί γιατί πρέπει να αξιολογείται αν είναι επικίνδυνοι ή επικίνδυνη η μαζική επεξεργασία των δεδομένων ουσιαστικά σχετίζεται με το πρόβλημα της εισαγωγής διακρίσεων, δηλαδή να αρνηθεί κάποιος την ευκαιρία ή να επιτρέψει σε ένα άτομο να μπει στη χώρα ανάλογα με την ε, εθνική ομάδα στην οποία ανήκει. Θέλετε να επαναλάβω τον ορισμό. Υπάρχει ούτως ή άλλως το κείμενο. No. Μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα για τους διερμηνείς. Και δυστυχώς χάνουμε τα μισά από ό,τι λέτε. Πρέπει να μιλάτε πιο αργά. Uh, Ζητώ συγγνώμη από τους διερμηνείς και από το κρατήριο. Όλα όσο έλεγα άλλωστε. Υπάρχουν στη μελέτη. Uh, υπάρχουν εδώ αντίγραφα. Οπότε μην τα για να ολοκληρώσω για τις συστάσεις. Αυτές οι συστάσεις ε, ουσιαστικά έχουν να κάνουν με το πώς πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις για το θέμα των ευφυών συνόρων και των βάσεων δεδομένων. Αυτό έχει να κάνει με την ε, ετήσια παρακολούθηση ε, δηλαδή υπάρχει ανάγκη υποβολής εκθέσεων σε τακτική βάση για όλες τις δραστηριότητες επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνουν χώρα σε σχέση με τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο στάδιο αυτό δεν έχουμε μια τέτοια ενοποιημένη επισκόπηση και ε, αυτό σίγουρα θα απαιτήσει συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων που έχουν πρόσβαση, καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες στην ίδια τους στη χώρα. Αυτή η υποβολή εκθέσεων θα ε, μπορέσει να επιτρέψει να ληφθούν από αποφάσεις για το αν θα συνεχιστούν τα εφιστάμενα συστήματα ή θα αναπτυχθούν καινούρια. Το πιο σημαντικά σημεία στη σύσταση, στη συστάση της μελέτης έχει να κάνει με τη δημιουργία προφίλ και με την αναγκαιότητα να αναπτυχθεί ένας νομικός ορισμός του profiling, της δημιουργίας προφίλ. Και συγκεκριμένα ποιο είδο δημιουργία προφίλ απαγορεύεται εντελώς και ποιο είναι ανεκτό και με ποια όρια. Αυτό θα πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια κυρίω, ε, καθώς ε, θα μιλάμε για ολοένα πιο αυτόματου ελέγχου στα σύνορα. Και Επίσης υπάρχει και το θέμα της προστασίας των δεδομένων ε, και το απορρίτου είναι ζωτικά αλλά όχι επαρκή. Η αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων εξορισμού θα πρέπει να συζητηθεί και κυρίως σε σχέση με τους συνεργειακούς ελέγχους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στην παρουσίαση της Κομισιόν για τις προτάσεις της περί των εξύπνων συνόρων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις αυτές που υποβάλαμε πριν από μερικές εβδομάδες. Καταρχήν γενικότερο στόχος της δέσμης αυτής είναι να εξυγχρονίσει και να ενδυναμώσει τον έλεγχο στα εξωτερικά μας σύνορα και ταυτόχρονα να καταστήσει τη διέλευσή τους ασφαλέστερη και απλούστερη. Και αυτό στα πλαίσια του ότι μόνο με υψηλή ασφάλεια στα εξωτερικά μας σύνορα μπορούμε να αποτολμήσουμε την πραγματική κατάργηση των εσωτερικών σύνορων. Θα σας περιγράψω τα διάφορα τμήματα της πρότασης ιδιαίτερα για τους ταξιδιώτες. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έρχονται για μικρή διαμονή την χάνουν της ίδιας μεταχείρισης, δηλαδή ελάχιστο αριθμό ελέγχων για τους ενωσιακούς και πλήρη έλεγχο για τους τρίτους. Υπάρχουν όμως και μερικές κατηγορίες που την χάνουν ιδιαίτερων διευκολύνσεων εκείνοι που ανήκουν στην κατηγορία των τοπικών μετακινήσεων. Για όλους τους υπόλοιπους είναι πλήρης ο έλεγχος. Και αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν κάποιος έρχεται στην Ευρώπη για πρώτη φορά ή για 25η. Αυτό ισχύει μέχρι τώρα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι λογικό, γιατί αυξάνονται οι ταξιδιωτικές ροές και έτσι αυξάνονται και οι ώρες, ο χρόνος αναμονής στα σύνορα και χρειάζονται και περισσότεροι φύλακες στα σύνορα των χωρών μας. Θέλουμε λοιπόν μία άλλη προσέγγιση που να επιτρέπει σε ορισμένα κατηγορίες ταξιδιωτών και ομάδων ταξιδιωτών μία πιο, έναν πιο διευκολυμένο, πιο εύκολο έλεγχο στα σύνορα. βασιζόμαστε σε μια διαδικασία προδιαλογής, προελέγχου, δηλαδή αυτούς που έρχονται συχνά ή αυτούς που μονίμως διαμένουν στην Ευρώπη οι ηθαγενείς οι πολίτες τρίτων χωρών να διευκολύνονται και να τη χάνουν ενός απλοποιημένου ελέγχου. Απλοποιημένος έλεγχος παρόμοιος με αυτόν που ισχύει και για τους ενωσιακούς πολίτες. Αυτό είναι ανάλογο με την κατηγορία θεωρήσεων, όπου ορισμένοι που ταξιδεύουν συχνά έχουν πολλαπλή θεώρηση, δεν χρειάζεται κάθε φορά να κάνουν αίτηση. Και μειώνει και το χρόνο αναμονή στα σύνορα, ενώ τώρα είτε έχετε απλή είτε πολλαπλή βίζα, γίνεται πάντα ο πλήρης έλεγχος. Χρειάζεται κάποιος έλεγχος στα σύνορα που να ξεχωρίζει τον κάποιον που έρχεται για μία φορά από κάποιον που έρχεται συνήθως. Το σύστημα αυτό ταύτισης των συνήθων ταξιδιωτών δεν εξαρτάται από την εθνικότητα του ξένου πολίτη. Ισχύει για πολίτες οποιασδήποτε χώρας εκτός Ευρώπης, ούτε εξαρτάται από οποιαδήποτε αμοιβαιότητα. Δηλαδή ένας πολίτης κάποιας τρίτης χώρας θα έχει πρόσβαση σε αυτό το σύστημα ανεξάρτητα από το αν οι ενωσιακοί πολίτες την κάτι ανάλογο στη χώρα του. Είναι λοιπόν έτσι καθολικό για να το πω έτσι. Και δείχνει ότι η προσέγγισή μας είναι προσωποκεντρική. Επιλέγουμε ορισμένους ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, δηλαδή ορισμένες κατηγορίες ταξιδιωτών. Επίσης χρησιμοποιούνται έτσι νέα εργαλεία για την απλοποίηση και επιτάχυνση των ελέγχων δηλαδή τον αυτομητοποιημένο έλεγχο συνόρων που κάνει την ίδια δουλειά με τον φύλακα. Αυτές οι θύρες, οι πύλες, οι αυτοματοποιημένες έχουν δοκιμαστεί. Προς στιγμήν χρησιμοποιούνται μόνο από ενωσιακούς πολίτες, γιατί όπως σας είπα μόνο οι ενωσιακοί πολίτες απολαμβάνουν αυτόν τον απλοποιημένων ελέγχων. Οι δοκιμές ήταν πολύ θετικές και αποδοτικές επιτρέπουν όντως λιγότερο χρόνο αναμονής και είναι ένα πιο ευέλικτο εργαλείο στη διαχείριση των ταξιδιωτικών ροών, των επιβατικών ροών ή ροών επιβατών. Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα και για εξωενωσιακούς πολίτες που ανήκουν στις κατηγορίες που ανέφερα. Αλλά δεν εξαρτάται το σύστημα από τις αυτόματες αυτές στήρες. Υπάρχουν και οι συνήθεις με φύλακες, αλλά πάλι με απλοποιημένο έλεγχο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα, αλλά αυτό εξαρτάται από τις χώρες μέλη, να χρησιμοποιούνται οι ίδιες, οι ίδιοι διάδρομοι και ουρές με τους ενωσιακούς πολίτες. Ως προς τις ομάδες στόχευσης, αυτό είναι πάντα το πιο δύσκολο, αναμένουμε περίπου 5 εκατομμύρια να ζητήσουν να υποφελθούν από αυτό το πρόγραμμα το χρόνο. Αυτό αρθριστικά διότι κανείς υποφελείται από το πρόγραμμα αυτό για 5 χρόνια. Αλλά πρέπει να προσθέσουμε σε αυτόν τον αριθμό και εκείνους που είναι μόνιμοι κάτοικοι στην Ένωση και μπορούν επίσης να υποφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα μερικά θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επιλέξαμε ένα σύστημα που συνδυάζει μία κάρτα με την κεντρική τράπεζα δεδομένων. Η χρησιμοποίηση αυτής της κάρτας μας επιτρέπει να διαχωρίσουμε τα βιομετρικά από τα υπόλοιπα στοιχεία. Έτσι πιστεύουμε ότι μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε όχι μόνο τη χρήση των βιομετρικών στοιχείων αλλά και την πιθανή χρήση των υπολείπων. Τέλος, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του συστήματος για λόγους αστυνομικών ελέγχων. δεύτερο στοιχείο του προγράμματος αυτού εξύπνων συνόρων. Όπως ξέρετε, ο κύριος κανόνας για τους εξωενωσιακούς πολίτες που έρχονται για μικρή διαμονή περιορίζεται σε τρίμηνη με εξάμηνη περίοδο. Σήμερα, ο μόνος τρόπος που έχουν τα κράτη-μέλη για να επιβάλλουν τον κανόνα αυτό ή για να, τον, για να επιτηρήσουν είναι το σφράγισμα του διαβατηρίου. Αυτό ισχύει σήμερα. Όλα τα διαβατήρια των εξωενωσιακών πρέπει να σφραγίζονται στην είσοδο και έξοδο κάποιας χώρας. Αυτό όπως έχουμε ξαναπεί είναι κάτι που δεν λειτουργεί πολύ καλά. Γιατί όσοι ταξιδεύουν συχνά γεμίζουν τα διαβατήριά τους με εκατοντάδες σφραγίδες που είναι και δυσανάγνωστες και δεν μπορούν να τις ελέγξουν ούτε οι φύλακες πολύ καλά για να καταλάβουν πόσος χώρος χρόνος παραμονής τους μένει. Αυτή η περίοδος τριών με έξι μηνών μέχρι στιγμής εξαρτάται απολύτως ο έλεγχός της από τη, από τη σφραγίδα. Η κατάργηση του σφραγίσματος θα μπορούσε να αντικατασταθεί με ηλεκτρονική καταγραφή των ημερομηνιών εισόδου και εξόδου των εξωενωσιακών τουριστών. Όσοι έρχονται για μακρύτερη παραμονή ή είναι μόνιμοι κάτοικοι στην Ένωση δεν θα τους επιβάλλεται αυτό το σύστημα ηλεκτρονικού σφραγίσματος εξόδων-εισόδων. Θα μπορεί όμως έτσι ο φύλακας των συνόρων να γνωρίζει πόσο χρόνο διαθέτει κάποιος για να παραμείνει σε ενωσιακή επικράτεια και η πληροφορία αυτή μπορεί να χρησιμεύει και στον ίδιο τον ταξιδιώτη. Σήμερα δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε στα σύνορα αν πει ο επιβάτης, ο ταξιδιώτης πόσες μέρες μου μένουν από την τρίμηνη άδειά μου δεν μπορεί να το απαντήσει ο φύλακας γιατί θα πρέπει να κάνει υπολογισμούς και να συμβουλευτεί 20 σφραγίδες. ενώ με το καινούργιο σύστημα θα γίνεται. Επίσης θα χορηγεί πληροφορίες για τις αρχές των κρατών για όσους δεν σέβονται τις περιόδους, που δεν φεύγουν δηλαδή από την περιοφέρεια του Σέγγεν μέσα στους 3 ή 6 μήνες που τους έχουν δοθεί. Μετά από μια μεταβατική περίοδο το σύστημα θα χρησιμοποιεί και βιομετρικά στοιχεία για την καλύτερη ταύτιση όσων έχουν εισέλθει στην επικράτεια αλλά έχουν χάσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα παραδείγματο χάρη. Η μεταβατική περίοδος βασίστηκε σε εκείνη που είχαμε προβλέψει και για τις θεωρήσεις ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν τον χρόνο να προσαρμοστούν, να μετεκπαιδεύσουν το προσωπικό τους κλπ. Μέχρι να συνηθίσουν στα βιομητρικά Θέματα προστασίας στοιχείων λοιπόν είναι πολύ βασικά εδώ. Ιδιαίτερο κάτι που εξετάσαμε πολύ προσεκτικά και πολύ χρόνο να γι' αυτό είναι η πρόσβαση στο σύστημα για λόγους επιβολής του νόμου και της τάξεως. θεωρούμε από μελέτες ότι θα μπορούσε το σύστημα να χρησιμοποιηθεί και για την καταπολέμηση σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, αλλά δεν νομίζουμε ότι σε αυτή τη φάση έχουμε επαρκή πληροφόρηση και δεδομένα στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτό το σύστημα θα ήταν αναλογικό και απαραίτητο και για αυτούς τους λόγους. Γι' αυτό η Κομισιόν δεν προβλέπει χρησιμοποίηση του συστήματος για λόγους ε, αστυνομικούς. Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας του συστήματος θα το ξαναδούμε και θα αξιολογήσουμε όχι μόνο πώς δουλεύει για τις εισόδους-εξόδους, αλλά και τι εμπειρίες θα υπάρχουν και από το σύστημα των θεωρήσεων και για αστυνομικούς λόγους. Και τότε θα δούμε αν χρειάζεται νέα πρόταση για παράταση του συστήματος και για αστυνομικούς λόγους. Άλλο θέμα προστασίας δεδομένων, η περίοδος κατακράτησης των στοιχείων ή αποθήκευσης. Κατ' εμάς ο ελάχιστος χρόνος είναι έξι μήνες, γιατί αυτό ανταποκρίνεται στις συνήθεις περιόδους ε, διαμονής που χορηγούνται σε όλους. Προτείνουμε λοιπόν να μην ξεπεράσουμε αυτό το διάστημα. Μετά από έξι μήνες τα στοιχεία θα διαγράφονται. Βέβαια πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις για όσους δεν έχουν φύγει από τη χώρα του Σέγγεν μέσα σε έξι μήνες αυτούς. Αυτονών τα στοιχεία θα κρατιούνται για πέντε χρόνια το πολύ. Και αν κάποιος δεν έχει ποτέ συλληφθεί η διαπράξη αδίκημα αλλά δεν έχει φύγει από το Σέγγεν πάλι πρέπει να υπάρχει ανώτατος χρόνος κατακράτησης και νομίζουμε ότι πρέπει να είναι πενταετής. Τέλος για το σύστημα εισοδεξόδων επίσης υπάρχει η δυνατότητα να μοιραστούμε, να χορηγήσουμε δεδομένα και σε τρίτες χώρες, πράγμα που ισχύει και για το σύστημα των θεωρήσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επιστροφής. Η σύνδεση των δύο συστημάτων τώρα. Υπάρχει μία πολύ σημαντική σύνδεση. Όπως είπαμε το σύστημα εισοδεξόδων επιτρέπει την κατάργηση των σφραγίσεων και άρα πλήρη αυτοματισμό. Άρα συνδέονται τα δύο συστήματα μεταξύ τους, δηλαδή το σύστημα ισοδεξόδων μας επιτρέπει να κάνουμε και ημιαυτοματοποιημένους ελέγχους για τους ταξιδιώτες που έχουν ήδη εγκριθεί η καταγραφή. Τέλος, από την τεχνική πλευρά, η ανάπτυξη των νέων συστημάτων θα ανατεθεί στη νέα υπηρεσία στο Τάλιν και χρησιμοποιούμε το ίδιο τεχνικό σύστημα, την ίδια πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε και για τις θεωρήσεις. Um, η διαφορά είναι ότι η εφαρμογή αυτών των νέων προτάσεων θα αρχίσει μόνο αφού εγκριθούν από τους συνομοθέτες πρώτον για να μην προδικάσουμε τις επιλογές που μπορεί να κάνουν άλλες επιλογές που μπορεί να κάνουν οι συνομοθέτε. Δεύτερον, για να είμαστε βέβαιοι ότι οι, τα, οι απαιτήσει για τα κριτήρια του συστήματος έχουν εγκριθεί πριν αρχίσει η τεχνική τους εφαρμογή. Και τέλος, το κόστος. Αυτά είναι πολύ ακριβά συστήματα. Προτείναμε για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας 1,1 δισεκατομμύρια και για τα δύο συστήματα. Πράγμα που καλύπτει όχι μόνο την ανάπτυξη του συστήματος αλλά και τη συντήρησή του για την πρώτη τρι, τριετή ή πενταετή περίοδο. Είναι δηλαδή με το κλειδί στο χέρι αυτό το κόστος που σας λέω. Εξετάσαμε όσο καλύτερα γινόταν το κόστος αυτό, συγκρίναμε και τις επιπτώσεις που θα είχε το κόστος αυτό στην κανονική του λειτουργία καθώς και σε περιπτώσεις τεχνικών δυσκολιών δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των διαφορών επιλογών τεχνικών επιλογών που να μας επιτρέπει να πούμε ότι η μία είναι πολύ φτηνότερη από την άλλη αλλά υπάρχουν εξοικονομήσεις με το συνδυασμό των δύο συστημάτων παράλληλα παράλληλη εφαρμογή. Επίσης πρέπει τη χρηματοδότηση να την ξαναδούμε ανάλογα με το ποια θα είναι η τελική απόφαση για το επόμενο Πολδίπ μόλις και αν εγκριθεί. Μπορεί να σας φαίνονται όλα αυτά πολύπλοκα και ακριβά, αλήθεια είναι αυτό, αλλά επίσης πρέπει να δούμε σε σύγκριση με το τι ισχύει τώρα στην περιφέρεια του Σέγγεν, στον χώρο του Σέγγεν, που αφορά περίπου 500 εκατομμύρια κατοίκους και έχει τεράστια σύνορα και εκατοντάδες διελεύσεις το χρόνο. Και αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να διαχειριστούμε τις ροές αυτές αποτελεσματικά, ότι πρέπει όντως είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε αυτά τα ακριβά συστήματα. Σας ευχαριστώ κύριε Νίλσον. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Πουταρέλη από το EDPS. Σας ευχαριστώ πρόεδρε και ασφαλώς σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε για να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση για το πακέτο για τα ΕΦΗ e σύνορα. Ο υπεύθυνο ε, για την δημοσιεύσει μας έχει μόλις ε, δημοσιεύσει ένα tweet και αναφέρεται ότι η DPS θα εγκρίνει σύντομα μία θέση βάσει της ανάγκης, της αναλογικότητας και της ανάγκης μιας προσέγγισης που θα προσανατολίζεται στις μελλοντικές εξελίξεις. Αυτά ουσιαστικά θα ήθελα να σας πω σήμερα. Αναλύουμε στην παρούσα φάση μετά τα σχόλια που δημοσιεύσαμε τον Αύγουστο του περσινού έτους. Ε, αναλύουμε λοιπόν τα στοιχεία αυτά από πλευράς και προστασία των δεδομένων αλλά και υπό την ευρύτερη προοπτική. Και φυσικά μελετούμε τις βάσεις δεδομένων της δικαιοσύνης και των εσωτερικών ε, υποθέσεων και ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανταλλαγή δεδομένων. Θα θέλαμε ωστόσο να σας ενθαρρύνουμε όλους σας να σκεφτείτε παραπάνω για το πώς η ανταλλαγή πληροφοριών και τα ευρύτερα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να αναπτυχθούν στο μέλλον. Χτες μου έκανε εντύπωση η ομιλία του κυρίου Κοέλιο, ιδιαίτερα όταν ανέφερε ότι κάθε νέα πρωτοβουλία στον τομέα αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε κάποιες πρώτερες σκέψεις με βάση το πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τα νομικά εργαλεία και τις βάσεις δεδομένων που ήδη υπάρχουν. Πρωτού ξεκινήσουμε νέες πρωτοβουλίες δηλαδή. Αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι ασφαλώς και το κόστος όχι μόνο στα χρήματα αλλά και στα δικαιώματα του ατόμου σε ό,τι αφορά την ιδιωτική σφαίρα τα θέματα αποδοτικότητας ε, για την δημόσια ασφάλεια και να λάβουμε υπόψη ότι οι δύο προτάσεις συνεπάγονται την επεξεργασία δεδομένων τεράστιου αριθμού ατόμων. Ο κύριος Νίλσεν τόνισε πως η προστασία δεδομένων ε, αναγνωρίζεται στην ε, μελέτη αντικτύπου και στην έκθεση. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι η ανάγκη για μια τεράστια συλλογή στοιχείων ε, μας κάνει να σκεφτούμε κάποια θέματα. Καταρχάς, το σύστημα εξόδου σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τα άτομα που παραμένουν και μετά τη λήξη της παραμονής τους, της νόμιμης παραμονής τους και ενδεχόμενες κυρώσεις. Ε, για παράδειγμα, η μελέτη αντικτύπου αναφέρει ότι πάρα πολλοί μετανάστες μένουν πέρα από το διάστημα της ε, νόμιμης διαμονής τους, παραμονής τους. Αλλά διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία σε ό,τι αφορά τους ε, τα άτομα που λαθρέα διαμένουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Μπορούμε να συλλέξουμε περαιτέρω πληροφορίες με ανώνυμα στοιχεία, για παράδειγμα. Είναι βασικό να αξιολογηθεί καλύτερα το θέμα της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Καταλαβαίνουμε και ε, ομολογούμε ότι υπάρχουν δυσκολίες σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για την ε, λαθρέα μετανάστευση. Και αυτό θα επηρέαζε ασφαλώς και τη μεταναστευτική πολιτική μας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε και να αντιλαμβανόμαστε ότι η ελλείψη τέτοιων αξιόπιστων στοιχείων τα μέτρα που παίρνουμε για να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα μπορεί να είναι δυσανάλογα ή μη αποτελεσματικά. Και κάθε παρέμβαση στα δικαιώματα του πολίτη θα πρέπει να βασίζεται σε αδιάσυστα στοιχεία σχετικά με την αναγκαιότητά τους. Άρα θα πρέπει να γίνει περαιτέρω ανάλυση για το πακέτο για τα σύνορα και πώς αυτό μπορεί να σχετίζεται και με άλλα προγράμματα και πώς μπορεί να επηρεάσει τους ταξιδιώτες σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την είσοδό του στο χώρο Σέγγεν. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί λοιπόν το άρθρο 96 της Σύμβασης Σέγγεν προκειμένου τα άτομα τα οποία γνωρίζουμε ότι θα παραμείνουν και πέρα από τη λήξη τη άντρε παραμονή του να μην ε, λαμβάνουν είσοδο στο χώρο Σέγγεν. Για τα βιομητρικά στοιχεία, οι νέε προτάσεις βασίζονται στη χρήση τέτοιων στοιχείων και αναγνωρίσαμε σε διάφορε περιπτώσει ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα. Υπάρχουν ορισμένα πλεονεκτήματα από τη χρήση βιομητρικών στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται αυστηρέ προδιαγραφέ και δικλείδε ασφαλεία. Τα αριθμητικά στοιχεία αποτελούν ένα πρώτο στοιχείο για τα βιομετρικά στοιχεία στην αιτιολογική σκέψη 8. Αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθούν τέτοια ε, αριθμητικά στοιχεία και μετά από κάποια χρονικά διαστήματα και αποτυπώματα. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, όπως οι υποχρεώσεις των κρατών μελών να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες και θεωρούμε ότι τα βιομετρικά στοιχεία θα πρέπει να θεωρούνται μόνο ε, πρόσθετα στοιχεία σε περίπτωση που τα αριθμητικά στοιχεία δεν αρκούν. Αυτό που καθίσατε σαφές είναι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την πρόταση σε ό,τι αφορά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος εισόδου-εξόδου θα πρέπει να περιλαμβάνει σχέσεις που θα λαμβάνουν υπόψη και άλλους παράγοντες. Είναι λοιπόν σημαντικό να τονίσουμε και να αναγνωρίσουμε ότι η μελέτη αντικτύπου θα πρέπει να ζυγίσει όλα τα εμπλεκόμενα συμφέροντα και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εύκολη δικαιολογία για την παρέμβαση των αρχών. Να προτείνουμε και μια διατύπωση που θα αποτιμώνει καλύτερα το σημείο αυτοκίνησης. Νομίζω ότι με τις εμπειρίες του παρελθόντος ξέρουμε ότι όπου χρειάζεται πρόσβαση των αρχών σε τέτοια δεδομένα σε ό,τι αφορά άτομα τα οποία δεν είναι ύποπτα αυτή η πρόσβαση θα πρέπει να εκτιμάται και να αξιολογείται με πολύ μεγάλη προσοχή. Διάφοροι έχουν ασκήσει κριτική σε ό,τι αφορά τις τάσεις αυτές. Άρα, με την ευκαιρία αυτή, να σας υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να αξιολογούνται πάντα τέτοιες προτάσεις και ότι η ανάλυση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε μια ομοιόμορφη ενιαία προσέγγιση για το ζήτημα αυτό. Η μεταφορά σε τρίτες χώρες των δεδομένων αποτελεί άλλο ένα θέμα το οποίο πρέπει προσεκτικά να το εξετάσουμε. Θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις οι οποίες θα πρέπει ενδεχομένως να αναδιατυπωθούν. Τα πρόγραμμα των ταξιδιωτών. Θα δημοσιεύσουμε το, την ομιλία μου, θα βρείτε κάποια σημεία όπου θεωρούμε ότι θα πρέπει να εστιαστούμε στις πρακτικές συνέπειες των νέων συστημάτων, όπως για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο διακριτικής μεταχείρισης, σε ό,τι αφορά τον χρόνο αναμονής στους ε, συνοριακούς ελέγχους. Όλα αυτά αναλύονται και με βάση τα προγράμματα εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερώσουμε για τις πτυχές αυτές. Συνοψίζοντας λοιπόν τα συστήματα αυτά δημιουργούν όλα μία επιπλέον επέμβαση αν θέλετε στα δικαιώματα του ατόμου και αυτό είναι θεμητό μόνο εφόσον είναι όχι μόνο απαραίτητο αλλά και αναλογικό σε μια δημοκρατική κοινωνία. Θα καταθέσουμε μια γνωμοδότηση αλλά στις 10 Απριλίου να σας πούμε ότι έχει διοργανωθεί στο DPS ένας γύρος ε, τραπέζης ε, από επιστήμονες. Θα αποστείλουμε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Είσαστε όλοι προσκεκλημένοι, ιδιαιτέρως ε, οι συγητές και οι βοηθοί τους. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θα επικεντρωθεί σε λεπτομέρειες και επίσης θα συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες από τα κρατημέλη όπου υπάρχουν εμπειρίες από τον τομέα αυτό και θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή για να προβούμε σε περαιτέρω ανάλυση πρωτού τελικά καταλήξουμε στην τελική μας γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρο, Να δώσω πρώτα το λόγο στους δύο εισηγητές πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Καταρχάς, λοιπόν, η κυρία Ρενατέ Ζόμαρ, η οποία είναι εισηγητή για το σύστημα εισόδου-εξόδου και μετά ο κύριος Έντρου που είναι εισηγητής για το πρόγραμμα καταχωρισμένων ταξιδιών. Η κυρία Σόμερ έχει καταρχά το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους πανελίστε για την παρουσίασή τους. Είναι απόλυτα σαφές θεωρώ ότι ένα σύγχρονο σύστημα για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων είναι κάτι το απαραίτητο. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα εισόδου-εξόδου και χρειαζόμαστε και ένα πρόγραμμα για τους ε, καταχωρισμένους ταξιδιώτες. Ως τώρα δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά συστήματα ενδείξεως για το πότε μπαίνει και βγαίνει κάποιος στο χώρο Σέγγεν και είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο, είπαν οι ομιλητές. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει. Δεδομένου επίσης του γεγονότος ότι ε, απελευθερώνεται διαρκώς το σύστημα θεωρήσεων με τρίτα κράτη. Και φυσικά θα πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε κατά πόσον οι διατάξεις για τις θεωρήσεις τηρούνται και κατά πόσον ε, οι τρίτοι υπήκοοι τρίτων χωρών παραμένουν, διαμένουν νόμιμα στην Ένωση. Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων θα πρέπει να ενημερωθεί βάσει των πρόσφατων τεχνολογικών εξέλιξεων. Όλοι και αυτό υπογραμμίστηκε άλλωστε, ότι αυξάνονται οι παραβιάσεις των εξωτερικών συνόρων Διακώς. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία θα επιταχυνθεί περαιτέρω δεδομένης και της ε, αυξανόμενης ε, παγκοσμιοποίησης η έλεγχη, λοιπόν θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο εύκολη, γρήγορη και αυτοματοποιημένη. Αυτό διευκολύνει όχι μόνο τους ταξιδιώτες, αλλά και εμάς. Και το τόνισε ο κ. Μπουταρέλη πριν από λίγο. Θα καταπολεμούσε καλύτερα και τη λαθρομετανάστευση. Οι προτάσεις για τα συστήματα εισόδου, εξόδου και για το RTP θεωρώ κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση αλλά η πραγματική προστιθέμενη αξία του συστήματος εισόδου-εξόδου θα ήταν και η πλήρης αξιοποίηση των δεδομένων αυτών. Αυτό τι θα σήμαινε σε τελική ανάλυση, ότι θα μπορούσαν να διατεθούν και στις αρχές ποινική δίωξης. Καλό είναι να σκεφτόμαστε ιδιαίτερα σε ότι η προστασία των δεδομένων μέχρι που θέλουμε να φτάσουμε, αλλά αν έχουμε τα δεδομένα αυτή, γιατί να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για τους κατάλληλους ε, σκοπούς. Και εδώ το θέμα δεν είναι ο μικροεγκληματίας, μιλάμε για την δίωξη οργανωμένου εγκλήματος. Και νομίζω ότι αυτό θα αποτελούσε μια πολύ καλή ευκαιρία για την υποστήριξη των σχετικών διοκτικών αρχών. Θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον το σύστημα θα έπρεπε να βασίζεται εξ αρχής πλήρως σε βιομετρικά στοιχεία. Ακούσαμε κάποιες αμφιβολίες που εκφράστηκαν, αλλά πιστεύω ότι πρόκειται για την μοναδική δυνατότητα για την σίγουρη ταυτοποίηση των ε, προσώπων. Γιατί τι θα κάνουμε αν τα άτομα αυτά, για παράδειγμα, αφού έχουν μπει σε μια χώρα, έχουν καταστρέψει το διαβατήριό του. Χρειαζόμαστε στην περίπτωση αυτή τα βιομητρικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για ένα πρόγραμμα καταχωρισμένων ταξιδιτών τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αποφάσισε την πρόταση για ένα σύστημα βάση token τέτοια στοιχεία σωστή η πρόταση, αλλά έχουμε κάποια ερωτηματικά. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το επιπρόσθετο κόστος, το επιπρόσθετο γραφειοκρατικό άχθος. Και φυσικά υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος απώλειας, ο κίνδυνος ε, παραχάραξης. δεν θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρονικό διαβατήριο, το τυποποιημένο διαβατήριο χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, συμβάσεις ε, και με τρίτες χώρες. Αυτό το διαβατήριο λοιπόν θα μπορούσε να λειτουργεί σαν token και έτσι να αποφύγουμε μια κάρτα με chip Για τα βιομετρικά στοιχεία θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσον τα αποτυπώματα υπαρκούν. Η Μήπως θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η ηλεκτρονική εικόνα του προσώπου, πως τα ηλεκτρονικά διαβατήρια. Δεν έχουμε και εμπειρίες με τα token και το ερώτημα λοιπόν είναι κατά πόσον ε, θα ήταν πραγματικά ε, αξιόπιστη η λύση, γιατί στην παρουσία δεν έχουμε χρήματα και δεν πρόκειται σύντομα αυτό να αλλάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε λοιπόν ε, τα χρήματα για τέτοια ακριβά πειράματα. Ένα άλλο θέμα, το οποίο μας βρίσκει λίγο αντίθετος ε, από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ό,τι αφορά και το, το αμερικανικό σύστημα ΕΣΤΑ, το ηλεκτρονικό σύστημα έγκρισης ε, εισόδου. Θα είχε νόημα ένα τέτοιο σύστημα στην Ευρώπη να κάνουν δηλαδή online καταχώρηση ταξιδιώτες πρωτού μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια πλήρως, ένα πλήρες, πλήρως ε, ψηφιοποιημένο σύστημα για την είσοδο των ταξιδιωτών. Αλλά είναι σημαντικό γιατί πάντα είμαι υπέρμαχος ε, της προστασίας των προσωπικών δικαιωμάτων και της ιδιωτικής σφαίρας Ähm, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των στοιχείων σε τρίτα κράτη, θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, γιατί είμαστε πολύ επικριτικοί σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά εδώ στην Επιτροπή και σε ό,τι αφορά φυσικά τα συστήματα που συζητιώνται για το ΕΦΗ σύνορα. Να ρωτήσω τον κύριο Μπουταρέλη αν υπάρχει πλήρης ε, ψηφιοποίηση των δεδομένων, πότε θα έχουμε αποτελέσματα. Γιατί αυτά ε, ενδεχομένως θα πρέπει να τα εντάξουμε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τέλος, θα ήθελα συνολικά να αναφέρω ότι οι προτάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι κάτι το οποίο καλωσορίζουμε. Είναι πραγματικά κατεπηγόντως απαραίτητες. Έχουμε καθυστερήσει ήδη και σίγουρα θα έχουν επιπρόσθετη αξία και για τους ταξιδιώτες και για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να τονίσω ότι σε τελική ανάλυση το σύστημα ευφυών συνόρων θα προάγει και θα καταστήσει πιο ασφαλή την ελεύθερη μετακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δώσει στους πολίτες μας ένα πιο έντονο αίσθημα ασφάλειας. Και αυτό αποτελεί πάντα ένα θέμα το οποίο θίγουν οι πολίτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριο Έντσιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες που είναι παρόντες εδώ. και φυσικά οι παρουσιάσεις τους μας βοηθούν να απαντήσουμε σε θέματα αρχής ε, για το σύστημα ευφυών συνόρων. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή πρέπει ακόμη να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε την πρόταση της Κομισιόν, κυρίως αν πιστεύουμε ότι, αν δούμε και τα δύο συστήματα ως καινοτόμα. Έχουμε μικρή εμπειρία για να κάνουμε συγκρίσεις. Το πιο σημαντικό θέμα, το πιο σημαντικό ερώτημα που θα πρέπει να θέσουμε έχει να κάνει με την αναγκαιότητα του να έχουμε αυτό το σύστημα ευφυών συνόρων και να ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά. Τα δέκα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει τα μάλα για να έχει ασφαλή σύνορα και να καταπολεμήσει την λαθρομετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε συστήματα βάση δεδομένων όπως το ΣΥΣ, το ΒΙΣ, το Eurodac και το Eurosur που αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση. Όμω, δυστυχώ, θα πρέπει να πω πω αυτέ οι προσπάθειε για την καταπολέμηση τη λαθρομετανάστευση δεν ε, συνοδεύονται και από μέτρα να ενθαρρύνουν την κινητικότητα στο χώρο Σέγγεν. Έχουμε όλο ένα και πιο δαπανερά συστήματα όπως το ΕΦΗ σύνορα φαινός, από είναι άλλη περιορίζουμε την κινητικότητα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ελεύθερη κυκλοφορία, την αναζήτηση εργασίας ή ε, μιλάμε για επαναθνικοποίηση του χώρου Σέγγεν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο, δηλαδή κινητικότητα και ασφάλεια, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε την κινητικότητα δίχω την ασφάλεια. Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε αυξημένη παρακολούθηση, εποπτεία και δημοκρατικό έλεγχο αυτή τη δομή και τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Τώρα βρισκόμαστε στο διακυβερνητικό στάδιο του χώρου Σέγγεν και δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν αρκεί. Πιστεύω λοιπόν ότι τα μέτρα παρακολούθησης των συνόρων και των ταξιδιωτικών ροών θα πρέπει να συνοδεύεται και από το μηχανισμό αξιολόγησης Σέγγεν ένα πολύπλοκο αρχιτεκτόνημα είναι άχρηστο αν δεν διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν σωστά τα συστήματα και γι' αυτό να σας πω ότι κατά την άποψή μου η πρόοδος που καταγράψαμε με αυτή τη δέσμη μέτρων για τα φυή σύνορα θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση του μηχανισμού Σέγγεν, από το μηχανισμό αξιολόγηση Σέγγεν. Τώρα θέλω να αναφερθώ στην ε, αναγκαιότητα για τα ευφύ σύνορα. Την λογικότητα. Πρέπει να θέσουμε το ερώτημα αν πραγματικά αποτελεί προτεραιότητα αυτό το σύστημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αλήθεια ότι προβλέπουμε μία σειρά ταξιδιωτών, μάλλον προβλέπουμε ότι ο αριθμός των ταξιδιωτών θα αυξηθεί και θα πρέπει να διευκολύνουμε τη διέλευση των συνόρων, αλλά θα πρέπει και να αναρωτηθούμε αν τα ευφυή σύνορα θα διευκολύνουν τη διέλευση των συνόρων ή αν θα την επιβραδύνουν τελικά. Σε ό,τι αφορά το σύστημα εισόδου-εξόδου, έχω την εντύπωση ότι θα αυξηθεί ο χρόνος αναμονής ε, στα μία διέλευση συνόρων, γιατί θα πρέπει στην είσοδο και στην έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίρνουν αποτυπώματα από όλου τους ταξιδιώτες και να δημιουργούμε και τεράστια αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα. Επίσης, άλλες καθυστερήσεις στα σύνορα θα οφείλονται στο ότι αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα δεν είναι αλάθητο, έτσι λοιπόν μπορεί να δημιουργηθούν λάθη. και σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Επίσης, θα πρέπει να σκεφτούμε και το επιχειρησιακό κόστος. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, πρόκειται για 1,1 δις ευρώ, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το κόστος των αυτόματων πυλών που θα πρέπει να πληρώσει το κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε αν σε αυτό το πλαίσιο τη οικονομική κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επενδύσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο σε τέτοια συστήματα ή αν αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλου σκοπού. Παίρνουμε χάρη για να έχουμε πιο ασφαλή ταξιδιωτικά έγγραφα ή breeder documents, έγγραφα πηγή. Θα πρέπει επίσης να εμβαθύνουμε και σε ένα άλλο ζήτημα, στο θέμα της χρησιμότητας του συστήματος εισόδου-εξόδου και του προγράμματος καταχωρημένων ταξιδιωτών. Εγώ δεν θα ήθελα τα εφή σύνορα ε, να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουμε μια νέα αστυνομία σύνορων πρέπει να μελετήσουμε το στόχο, το σκοπό αυτού του συστήματος. Θέλουμε να ελέγξουμε τη λαθρομετανάστευση, αλλά θα πρέπει να υπερισχύει ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα την καταχώρηση των ταξιδιωτών, νομίζω ότι είναι καλή η πρόταση της Κομισιόν. Βασίζεται στο προηγούμενο κανονισμό VIS-SIS, όμως υπάρχουν πτυχές που πρέπει να αποσαφινιστούν και θα αναφέρω ορισμένες. Παραδείγματο χάρη, η σχέση που θα έχετε το με τα, τα R2P, με άλλα συστήματα και με την αρχιτεκτονική του ΣΥΣ και του ΒΙΣ και με το σύστημα εισόδου-εξόδου. Επίσης, ε, για το πρόγραμμα καταχωρημένων ταξιδιωτών, νομίζω ότι δεν έχουν εκπονηθεί όπως πρέπει τα κριτήρια και οι αρμόδιες αρχές έχουν πάρα πολλές ελευθερίες. Ένα άλλο σημαντικό θέμα έχει να κάνει με την αξιοπιστία των ε, ψηφιακών αποτυπωμάτων και τη συλλογή του. Σκέφτομαι κυρίω τι ειδικέ κατηγορίε ανθρώπων, όπω είναι τα παιδιά και ηλικιωμένοι, αλλά και τα άτομα με αναπηρία. Το πιο σημαντικό πρόβλημα έχει να κάνει με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη χρήση τους κτλ. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, καθώς ο κύριος Μπουταρέλη παρουσίασε πάρα πολύ καλά τις ανησυχίες που υπάρχουν, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένες πτυχές πάρα πολύ σημαντικές. Σε ό,τι αφορά τις αρχές της αναλογικότητας. Δεν καταλαβαίνω σε τι χρησιμεύει στο να υπάρχει αντίγραφο ε, των εγγεγραμμένων ταξιδιωτών, καθώς υπάρχει κεντρική βάση δεδομένων, στην οποία έχουν πρόσβαση όλες οι αρχέ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πού είναι το νόημα να έχουμε δύο φορές τα δεδομένα αυτά και στην Εθνική Βάση Δεδομένων δηλαδή. Επίση, όταν ανακαλεί ένα άτομο το αίτημά του, θα έπρεπε να διαγράφονται αυτά τα δεδομένα, όχι να διατηρούνται για πέντε έτη όπω προτείνει η Κομισιόν. Επίσης, ε, θέλω να δηλώσω την ικανοποίησή μου που τα δεδομένα στο πρόγραμμα αυτό δεν μπορούν να διαβιβαστούν προς άλλα κράτη, προς διεθνείς οργανισμούς. Νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε την ίδια αρχή και για το σύστημα εισόδου-εξόδου. Ω προ την ασφάλεια των δεδομένων, νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερου τεχνικού συμβόλου ε, από την έννοια, παραδείγματο χάρη. Αυτά είναι ορισμένα στοιχεία προβληματισμού που ήθελα να σας παρουσιάσω σήμερα. Και όπως σας είπα, παραμένουν πάρα πολλά ζητήματα, υπάρχουν περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντήσεις. Και πιστεύω ότι για το επόμενο διάστημα θα ήθελα να συζητήσω με την κυρία Ζόμερ για να ε, μπούμε και σε συζήτηση και με την υπηρεσία του Τάλιν, με την Κομισιόν, με τους συναδέλφους, ε, με τους και εισηγητές και κλείνοντας να πω ότι η υιοθέτηση ενό αποτελεσματικού μηχανισμού αξιολόγηση έγκεν αποτελεί απαραίτητη προπόθεση για να σημειώσουμε πρόοδο σε ό,τι αφορά τα ευφυή σύνορα. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα ακούσει το μήνυμά μου και θα έχει μια επικοδομητική στάση για να μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε συμβεσμό σε αυτό το πακέτο Σέγγεν. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε και ποια είναι τα διδάγματα του παρελθόντος το χάρη, έχω κατά νου το σύστημα sis 2 και Eurosur. Πρέπει να έχουμε μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των ευφυών συνόρων. Ταυτόχρονα, κανένα πρόγραμμα εισόδου-εξόδου ή εγγεγραμμένων τοξιδιτών δεν θα πρέπει να ξεκινήσει πριν από την υιοθέτηση του κανονισμού από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Έντσιου. Τέσσερις συζήτησαν το λόγο. Έχω και εγώ μερικά σχόλια. Κανείς άλλος, ο κύριος Μπρόνς. Ο κύριος Ζάντε μίλησε για επιτρεπτά και μη επιτρεπτά στοιχεία κατηγορίες. Το profiling όμως νομίζω αυτού του είδους δεν είναι καθόλου λογικό. Οποιαδήποτε ομάδα από οποιαδήποτε χώρα μπορεί να εκπροσωπείται δυσανάλογα σε εγκληματικές δραστηριότητες. Επομένως δεν πρέπει να απαγορεύεται το profiling. Αν ας πούμε διαπιστωθεί ότι διδάσκαλοι γίνονται ευρωβουλευτές και μετά δουλέμποροι, οι κυρίες της μέσης τάξης στην Αγγλία καταλήγουν τρομοκράτες και πάντοτε το υποψιαζόμουν αυτό, τότε οι ομάδες αυτές πρέπει να χαρακτηρίζονται και να υποβάλλονται σε πληρέστερους ελέγχους και ανακρίσεις. Πριν από μερικά χρόνια για την εμπορία ανθρώπων εδώ μέσα είχα ρωτήσει ταπεινά τον εκπρόσωπο της Ευρωπόλ αν υπήρχε καμία ιδιαίτερη ομάδα του πληθυσμού που να εκπροσωπείται δυσανάλογα στους δουλεμπόρους ή στα θύματα αυτών και απάντησε όχι με τόση ταπεινότητα ότι δεν φταίγανε την κάνει και για τα δύο. Νομίζω ότι η μόνη ομάδα που υπερεκπροσωπείται εδώ μέσα κύριε Μπρόνς είναι αφορά τα φύλλα. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές. Λυπάμαι που έχασα μερικές ή περισσότερες από τις παρουσιάσεις σας γιατί είχα ψηφοφορία σε άλλη ή άλλες επιτροπές. Ό,τι άκουσα όμως ήταν πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό αν επαναλάβω κάτι που το είπαν άλλοι παρακαλώ να με συγχωρήσετε ή που είπατε εσείς μάλλον. Θα ήθελα να ρωτήσω για το κόστος κυρίως Ακούω κρίσης ότι είναι ψηλό το κόστος. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά διότι ήδη τώρα έχουμε προβλήματα με το Πολδίπ και το Συμβούλιο ζητάει περικοπάς. Και αν τα ευφυή στοιχήσουν έστω και το 1 τέταρτο του ISF, πρέπει να δούμε ποια είναι η προτεραιότητα. Είναι προτεραιότητα τα FEE e σύνορα και αν περικο... υπάρξουν περικοπές σε άλλους τομείς για να πληρωθεί αυτό, από πού θα γίνουν οι περικοπές, γιατί από κάπου πρέπει να προέλθουν τα χρήματα ή μήπω θα τα δώσουν τα κράτη-μέλη. Δεν νομίζω γιατί δεν θέλουν ούτε δεκάρα παραπάνω να δώσουν στο πολιτήφ. Πολδίπ. τι γίνεται και στην Κύπρο και αλλού. Μπορούν αυτοί να δώσουν περισσότερα χρήματα για έλεγχο στα σύνορα. ποιο θα παραμείνει σε αυτό το ύψος 1,1 δις. Αυτό ε, υπολογίστηκε στην πρώτη ανακοίνωση της Κομισιόν. Είχε ανακοινωθεί χαμηλότερο και ήδη αυξήθηκε. Ξέρουμε ότι είναι εύκολο να αυξηθεί το κόστος αφού μιλάμε για τεχνολογία και τις εξελίξεις της. Αναρωτιέμαι λοιπόν από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά. Εμείς ως Επιτροπή είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε περικοπές σε άλλους τομείς για να πληρώσουμε τα ευφυή σύνορα. Θα ήθελα να μου απαντήσουν και οι συνάδελφοι. Τώρα προς την Κομισιόν θα ήθελα να ρωτήσω και λυπάμαι αν το έχετε ήδη ξαναπεί, συγγνώμη. Αν διαπιστώσουμε ότι κάποιος παραμένει στο Σέγγεν περισσότερο χρόνο από ό,τι του επιτρεπόταν, τι θα γίνει. τι εφαρμόζεται νομικά. Θα ήθελα να ξέρω όλες τις λεπτομέρειες, αφού διαπιστώσουμε ότι κάποιος έχει ξεπεράσει το χρόνο διαμονής του, τι γίνεται. Ας σταματήσω εδώ, αν και είχα κι άλλα να πω για το σκοπό, τον ίδιο το σκοπό της συλλογή αυτών των στατιστικών στιγμών που θα είναι και πολύ ακριβώς. Ernst. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσω θα ήθελα καταρχάς ε, να απορρίψω και να πω ότι είμαι αντίθετη με αυτά που αναφέρθηκαν, γιατί νομίζω ότι αν ξεκινάμε έτσι, νομίζω ότι αποκρομακρυνόμαστε από κάποιες αρχές που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το θέμα τώρα το που μας απασχολεί. Να ξεκινήσω και εγώ για το θέμα, με το θέμα του κόστους. Κοιτώντας τι γίνεται στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θέμα του ΣΥΣ 2, θεωρώ ότι ήμουν πριν από δέκα χρόνια ε, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο όταν ε, συζητήθηκε το ζήτημα αυτό και αναφέρθηκε το θέμα του κόστους. Τώρα προστίθεται κι άλλους και προστίθεται και άλλα συστήματα που κοστίζουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι κατά πόσον οι πόροι μπορούν να διατεθούν, όπως ρώτησε η κυρία Κέλλερ. Και για το 1,1 δισεκατομμύρια μπορεί να παραμείνει αυτό. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει κάτω, κάτι τέτοιο. Και θα πρέπει να δούμε τι μέσα διατίθενται για τη συλλογή τέτοιων δεδομένων και τι σκοπό εξυπηρετούν τα συστήματα αυτά και τι σκοπό εξυπηρετεί να δημιουργηθεί ένα καινούριο σύστημα που κοστίζει τόσο πολλά χρήματα με τόσε πολλέ χώρε. Το θέμα του κόστου, δηλαδή, καταρχά. θα ήθελα οι πανελίστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα απαντήσουν. Δεύτερο πρόβλημα. Η καταχώρηση. Έχουμε ένα πρόγραμμα καταχωρήσεω για του ταξιδιώτε πρώτη τάξεως και δεύτερη τάξεως. Έτσι το ερμηνεύω εγώ. Αυτό προκύπτει τα διάφορα κριτήρια. Το ερώτημα λοιπόν είναι σε τι μας ωφελεί. Όχι μόνο οι ταξιδιώτες, σε τι ωφελούνται, αλλά τι ωφελείται, σε τι ωφελείται και αυτός που κάνει την καταχώρηση. Οι επιχειρηματίες, για παράδειγμα, οι πολιτικοί αποτελούν χαμηλότερο παράγοντα κινδύνου. Οι άλλες κατηγορίες ε, ταξιδιωτών ε, παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο. Θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί να επιτρέπεται. Αλλά πιστεύω και πείτε μου και εσείς τι θεωρείτε ότι τα θέματα ασφάλειας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο εδώ. Για τον έλεγχο, για την εφαρμογή μηχανισμών ασφαλείας και ότι αυτός είναι ο στόχος και να περάσουμε στο σύστημα το θαυμάσιο εισόδου-εξόδου. Μας είπατε ότι καταργείται η σφραγίδα. Πολύ ωραία. Λιγότερες σφραγίδες, λοιπόν, στα σχετικά έγγραφα. Αυτό πολύ θετικό. Αλλά τι γίνεται. Κάποιος μπαίνει, βγαίνει, τον καταχωρίζω. Πρόκειται για ένα θέμα συγκεκαλυμμένης στατιστικής ε, μετανάστευσης. Δεν θεωρώ ότι μπορούμε να το ερμηνεύσουμε διαφορετικά αυτό που είπε η κυρία Κέλλερ, να ρωτήσω κι εγώ. Τι συμβαίνει μετά από τους τρεις μήνες, αν δεν έχει βγει το ταξιδιώτης. Θα εξαπολύσουμε τα σκυλιά να βγουν, να ψάξουν το άτομο που έχει μείνει μέσα στην επικράτεια της Ένωσης. Τι θα συμβαίνει, τι θα συμβεί. Υπάρχει κάποια ρύθμιση. Και τώρα για τα βιομετρικά στοιχεία είναι ανοησία ότι τα βιομετρικά στοιχεία, τα οποία προστίφονται στα στοιχεία που ήδη περιλαμβάνονται στα συστήματα, δεν είναι καθόλου ασφαλή αυτά τα βιομετρικά στοιχεία, να σας πω και να σας θυμίσω το χάος που είχε προκύψει όταν αποκαλύφθηκε πόσο εύκολο ήταν γίνει νοθεία σε αυτά τα βιομετρικά στοιχεία μέσω υπολογιστή. Άρα αυτό πραγματικά είναι ανοησία αυτή η αιμονή στα βιομετρικά στοιχεία. Και έτσι λοιπόν ερωτώ στην τελική ανάλυση ποιος τελικά ωφελείται ο ταξιδιώτης λόγω της φραγίδας. Τι να σας πω, αμφιβάλλω, θεωρώ ότι καταλήγουμε σε θέματα πολιτικής ασφάλειας. Και όταν αρχίσουμε να εξετάζουμε τέτοια θέματα, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το θέμα της υπηκότητας. Ο κύριος Τόρβαλς. Ευχαριστώ. Άκουσα τη συζήτηση και όταν κάνουμε τέτοιε συζητήσει, σχεδόν πάντα φοβάμαι ότι επικεντρωνόμαστε στα λάθο πράγματα. Ποια είναι τα κυρία ζητήματα με το όλο πακέτο, είναι Δηλαδή, σε σχέση με τις διελεύσεις ε, των σύνορων, ε, τι θα γίνει ε, στο μέλλον, θα έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό διελεύσεων. Ο στόχος είναι να συλλάβουμε όσους μένουν παραπάνω παρανόμως ή να συλλάβουμε όσους δραστηριοποιούνται στο οργανωμένο έγκλημα. Επομένω, αν δούμε τα αριθμητικά στοιχεία, πόσες διελεύσεις ε, σύνορων έχουμε και πόσους θα έχουμε που θα μένουν παραπάνω παρανόμω και πόσους ε, δράστες ε, σοβαρών εγκλημάτων θα πιάσουμε με το σύστημα αυτό. Φοβάμαι ότι θα μιλήσουμε για εκατομμύρια διελεύσεις σύνορων και για εκατοντάδες ή χιλιάδες, ίσως ένα εκατομμύριο ατόμων που θα διαμένουν παραπάνω παράνομα. Πρέπει να δούμε τις αναλογίες και αν δεν δούμε αυτές τις αναλογίες... Κάποιοι θα μιλούν ε, για το ένα και κάποιοι για το άλλο, για άσχετα πράγματα δηλαδή. Και έχουμε και το θέμα του κόστους. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να φοβούνται την αύξηση του κόστους. Τουλάχιστον στη δική μου χώρα, τουλάχιστον κάθε πρόγραμμα που αφορά την αποθήκευση δεδομένων, ε, για κάθε πρόγραμμα δεφανήθηκαν τρομερά ποσά. Και όσοι προσπαθούν να μας πουλήσουν τέτοια προγράμματα, Μα λένε συνήθως ότι θα είναι μικρό το ποσό και μετά από 10 χρόνια τελικά βλέπουμε ότι αυτό το ποσό δεν ήταν και τόσο μικρό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να είμαστε ειλικρινεί εδώ σε σχέση με το θέμα του κόστου. Και ρώτησα και νωρίτερα στη συζήτηση ποια αρχιτεκτονική χρησιμοποιούμε, δηλαδή δημιουργούμε νέα προγράμματα για, σε, πάνω σε ξεχωριστές νέες πλατφόρμες και η απάντηση που πήρα είναι ότι αυτό δεν είναι ένα κανονικό πρόγραμμα. Είναι ουσιαστικά μια νέα πλατφόρμα που θα οικοδομηθεί αποκλειστικά για αυτό το πρόγραμμα και τι το καλό θα την κάνουμε. Δηλαδή κάνουμε κάτι με συνηθισμένα building blocks, με συγκεκριμένα στοιχεία ή εδώ εφεύρουμε κάτι καινούριο για την ίωστη φορά. Επομένως, δεν ήθελα να ακούσω ποια είναι τα κύρια οικοδομικά στοιχεία εδώ, πώς συντεριάζονται και τι είδους πρόγραμμα τελικά χρησιμοποιούμε. Δηλαδή θα έχουμε μια πλατφόρμα που θα βασίσει στα Windows, μια πλατφόρμα Linux, τι πλατφόρμα έχουμε τελικά. Σε ποια πλατφόρμα θα τρέχει το πρόγραμμα. Ε, πώς ε, θα μπορεί να επικοινωνεί αυτή η πλατφόρμα με τα νέα στοιχεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοέλιο, τελευταίος ομιλητής πριν από μένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία ζητήματα. Προτεραιότητα, το θέμα της προτεραιότητας, ε, το θέμα του κόστους και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, σύνδεση με άλλα θέματα. Καταρχήν το θέμα των προτεραιοτήτων. Αυτό αναφέρθηκε από τους ομιλητές. Να είμαστε εντελώ ξεκάθαροι. Εμείς ε, δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι κρηματοοικονομικοί προορισμοί για τα επόμενα 7 χρόνια. Δεν γνωρίζουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές. Παρουσιάστηκαν ε, βέβαια αυτές οι δημοσιονομικές προοπτικές και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται να μας προτείνει μία επένδυση τέτοιου είδους, εγώ θεωρώ ότι είναι λογικό και σοβαρό να ρωτήσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες. Αυτό κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, να μας πει ποια είναι τα προγράμματα που θα υποτιμηθούν ή θα ξεχαστούν, γιατί φυσικά δεν θα υπάρχουν χρήματα για όλα και από πολιτική σκοπιά εμείς θα μπορούσαμε να πούμε αυτό είναι προτεραιότητα, όμως σίγουρα υπάρχει κάτι που μέχρι τώρα ήταν προτεραιότητα και θα πάψει να είναι. Αυτή η πολιτική μετάφραση πρέπει να γίνει. Αν η Ευρωπαϊκή πολιτική Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό είναι προτεραιότητα, πρέπει να μας πει τι θα πάψει να είναι προτεραιότητα. Επίσης, σε θέση με το οικονομικό κόστος και πόσο θα αποκλίνουμε τελικά το ΣΥΣ, ξεκίνησε με πρόβλεψη 25 εκατομμύρια ευρώ ξεχνώντας αυτά που δόθηκαν στα κρατη για να τα βοηθήσουν με τις εθνικές δαπάνες. Μιλάμε εδώ ε, για 260 εκατομμύρια ευρώ το 2012. Αν εμείς κάνουμε το ίδιο λίστημα και για το project αυτό, δηλαδή το 1,1 δις που προβλέπονται, θα μπορούσε να φτάσει στα 7 ή στα 8 δισεκατομμύρια στο τέλος του προγράμματος. Μπορείτε να πείτε ότι υπερβάλλω, ίσως, αλλά να λάβετε υπόψη και τη συνέβη στο παρελθόν, στο πραγματικό παράδειγμα του παρελθόντος. Και αυτή η διάσταση οικονομική δεν μπορεί παρά να μας ανησυχεί πραγματικά. Και τέλος, κάτι που υπόθηκε και από τον συνάδελφο Έντσιου, το θέμα της σύνδεσης με άλλα θέματα. Προβλέπεται να υπάρχει μια τεχνική πλατφόρμα, να βασιστεί στη τεχνική πλατφόρμα του ΣΥΣ, το ΣΥΣ δεν λειτουργεί. Θα λειτουργήσει, αλλά θα χρειαστεί μια περίοδο δοκιμών και προσαρμογή. Αν εγώ κατάλαβα καλά αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ε, πρώτη συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί, το ΒΙΣ θα είναι πλήρως επιχειρησιακό μέσα σε δύο χρόνια όλες οι συνδάσεις με τα υφιστάμενα συστήματα θα πρέπει να τις σκεφτούμε όχι μόνο από τεχνολογική σκοπιά, αλλά και για να αποφύγουμε την δημιουργία διπλών μέσων. Δηλαδή να μην αναζητούμε απαντήσεις που ήδη εν μέρη μπορεί να έχουν δοθεί από τα ισχύοντα συστήματα. Και για να κλείσω, Πρόεδρε, και για θέματα προτεραιότητας που δεν μου φαίνονται προφανείς αυτή τη στιγμή, είτε για λόγους ε, οικονομικούς, είτε για λόγους σύνδεσης με τα φυστάμενα συστήματα, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πολύ σόφρονες απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία πάρα πολύ σόφρονες. Εδώ, αν βιαστούμε, θα είναι μοιραίο κυρίως αν αυτό που θα μας οθήσει θα είναι η πολιτική της ασφάλειας. Όλοι είμαστε υπέρ της ασφάλειας, αλλά εδώ το μέτρο της αναλογίας είναι ουσιαστικό και πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά πολύ σοβαρά. Σας ευχαριστώ. Yes, thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο. Αν δεν θέλει κανείς άλλος, δεν έχω δει κανέναν να ζητάει το λόγο, θα σχολιάσω εγώ. Θα θέσω μερικά ερωτήματα στον κύριο Νίλσεν της Εκοκομισιόν. Αν ήμουν νεογέννητο, μπορεί να θεωρούσα και πολύ πιστική την πρότασή σας. Αλλά δεν είναι η πρώτη τέτοιο είδους πρόταση και όλοι μας εδώ Θέσαμε ερωτήματα για το κόστος. Μπορώ να σας δώσω κατάλογο όλων των μεγάλων πληροφορικών προγραμμάτων σε όλους τους προϋπολογισμούς και θα δείτε τι σύγκριση θα γίνει για το κόστος. Υπάρχουν παραδείγματα προς μίμηση. Ε, Ηνωμένε Πολιτεία, ας πούμε, προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο αυτοματοποιημένο σύστημα εισοδεξόδων, αλλά από ό,τι ξέρω και μετά από χρόνια δεν είναι ακόμη πλήρως λειτουργικό. Αν οι Αμερικανοί δεν μπορούν να τα καταφέρουν, γιατί να μπορέσουμε εμείς. Το κύριο ερώτημα το έθεσε ο κύριος Τόρβαλτ. Ποιος είναι ο στόχος. Είναι όπως είπατε να επιταχυνθεί η διέλευση των συνόρων. Τότε θα σας έλεγα το ίδιο, θα το πίστευα αν ήμουν προτάρα, αλλά Πόσα μέτρα έχουν περάσει από την Επιτροπή που μας έλεγαν ότι όλα αυτά θα αποσυμφορήσουν τα, τις ουρές στα αεροδρόμια. Έχετε δει εσείς καμία κατάργηση ουρών στα αεροδρόμια, εγώ δεν έχω δει. Μετά μίλησαν για σκάνερ σωματικά και κτλ. Δεν γίνονται όλα αυτά. Ε, ποιος είναι ο πραγματικός στόχος λοιπόν. Μήπως να συλλάβουμε πιο εύκολα όσους παραβιάζουν την περίοδο παραμονής. Αυτό γίνεται και με άλλες μεθόδους. Και από τα κινητά τους γίνεται. Και η αστυνομία τα έχει τα στοιχεία. Λοιπόν, ως προς την πρόσβαση για αστυνομικούς λόγους, πάλι αν ήμουν προτάρα θα πίστευα την υπόσχεσή σας ότι οι αστυνομικές αρχές δεν θα έχουν πρόσβαση. Πρέπει να σας πω για το Eurodac τι έγινε. Τι αξία έχει μια υπόσχεση της Κομισιόν. Γιατί εγώ να δεχτώ κάτι που αποδείχτηκε ότι δεν θα το εφαρμόσει η Κομισιόν. Γιατί να δώσω εμπιστοσύνη στην Κομισιόν. Για τις τράπεζες δεδομένων. Εκτός από την ασφάλεια που πρέπει να έχουν. Έχετε καθόλου σκεφτεί ποιος θα διαχειριστεί τα συστήματα και τις τράπεζες δεδομένων στους κανόνες που ισχύουν στον ΠΟΕ. Μπορούμε να ζητήσουμε να μην γίνεται η διαχείριση με βάση το Patriot Act, δηλαδή ότι θα είναι καθαρά ευρωπαϊκή υπηρεσία και δεν θα δίνει πρόσβαση σε άλλες κυβερνήσεις. Εκτός αν αποφασίσουμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα, αλλά αν υπάρχει μια εταιρεία που έχει παρουσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτόματα θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα οι κυβερνητικές αρχές. Τέλος. Πάλι για το στόχο. Είναι και αυτό ένα θέμα ασφαλείας όπως είπατε, αλλά έχουμε, κάνει, έχουμε πάρει τόσα πολλά μέτρα για την ασφάλεια. Είμαστε ασφαλέστεροι. Επενδύσαμε πολλά λεφτά και δεν θα εξηγήσει βέβαια όπως είπατε 1,1 δισεκατομμύρια, αλλά πολύ πολύ περισσότερα, μην είμαστε αφελείς. Πόσο περισσότερη ασφάλεια θέλ, αγοράζουμε με αυτά τα χρήματα. Shall we take the, can we take the Μήπως μπορείτε να απαντήσετε με τη σειρά που έθεσαν τα ερωτήματα οι συνάδελφοι. Ωραία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα γενικό σχόλιο θα ήθελα να κάνω σε ό,τι αφορά την ιδέα ότι τα συστήματα είναι απολύτως απαραίτητα γιατί προστατεύουν τον πολίτη. Και εδώ νομίζω ότι μπαίνει ερωτηματικό, γιατί ο κ. Νίλθεν είπε πολύ καλά ότι η ιδέα των ευφυών συνόρων έχουν να κάνουν ξεκινάνε από μια προσοκεντρική προσέγγιση. Το πρόβλημα είναι ότι αν ξεκινήσουμε με την προσέγγιση αυτή δεν ισχύει διάκριση μεταξύ πολιτών και παρανόμων λαθρομεταναστών. Γιατί αν ε, όλοι οι ταξιδιώτες καταστούν πιο επικίνδυνοι ή όχι εν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγχεται και ο χώρος που προστατεύεται. Αυτό έχει πολύ σημαντικές νομικές επιπτώσεις. Ε, άρα, τι ελεύθερη μετακίνηση μπορεί να υπάρχει όταν χρειάζεται επεξεργασία των δεδομένων και εξακολουθεί να ισχύει αυτή η ελεύθερη μετακίνηση υπονομικής άποψης. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίλης έχει το λόγο. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ και για τα πρώτα σχόλια που κάνετε για την προτάση αυτή που αποτελεί την αρχή μιας μακράς διαδικασίας και εντελεχούς διαδικασίας. Θα πρέπει να εξεταστεί από τα θεσμικά όργανα με ε, προσοχή. Να σας πω τώρα κάποια πράγματα. Να κάνω την μπορώ δηλαδή, γιατί δεν έχω λεπτομερέστατες τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν. Καταρχάς για το σύστημα εισόδου-εξόδου και το σκόπο που εξυπηρετεί. Όντως, αυτό που προτείναμε ο σκοπός είναι να είναι, υπάρχει καλύτερη διαχείριση των συνόρων, καλύτερη διαχείριση του σεβασμού των διαδάξεων για σύντομες παραμονές. Και αυτό σημαίνει ότι στην ε, παρούσα φάση ε, ο σκοπός δεν καλύπτει την καταπολέμηση του εγκλήματος. Αυτή ήταν η επιλογή που κάναμε, αλλά εξαρτάται και από τον συνομοθέτη να μας πει τι πιστεύει να τονίσω εκ νέου ότι σε ό,τι αφορά θέματα αναγκαιότητας θα πρέπει να κοιτάξουμε την, ε, τον κανόνα των 3 έως 6 μηνών παραμονής. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ο νόμος αυτός ή όχι. Αυτό θεωρώ ότι αποτελείται βασικότερο θέμα που καλούμαστε να απαντήσουμε. Τι κάνουμε για τα άτομα που δεν σέβονται την διάρκεια παραμονής τους θα στέλνετε μια προειδοποίηση σε όλα τα κρατη σε ό,τι αφορά θέματα μετανάστευσης και έτσι θα υπάρχει μια επιπλέον πηγή πληροφοριών για τις αρχές αυτές όταν προσπαθούν να εντοπίσουν και να ε, πιάσουν τέτοιους, τέτοια άτομα. Αλλά δεν ε, πηγαίνουμε πέρα από αυτό. Αυτό εντάσσεται στο ήδη φυστάμενο νομικό πλαίσιο των κρατών μελών βάσει τη οδηγία ε, για τις επιστροφές που δίνει στα καρτιμέλη μια σαφή επιλογή όσοι δεν έχουν ε, δικαίωμα να παραμείνουν είτε θα, θα πρέπει να λάβουν το δικαίωμα αυτό είτε θα πρέπει να επιστραφούν. Άρα υπό την έννοια αυτή αποτελεί το σύστημα αυτό εισόδου-εξόδου ένα επιπλέον εργαλείο το οποίο όμως δεν τροποποιεί την υφιστάμενη νομική βάση το σκοπός του προγράμματος καταχωρισμένων ταξιδιωτών. Εξαρτάται από το πώς ε, τα βλέπουμε τα πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι ε, διαχωρίζουμε τον κόσμο σε επίπεδα κινδύνου. Θα έλεγα ότι μας επιτρέπει να διακρίνουμε μεταξύ εκείνων που έχουν χαμηλό κίνδυνο ή εκείνων που έχουν άγνωστο κίνδυνο. Γιατί όλοι όσοι έρχονται από άλλες ε, χώρες ε, αποτελούν ένα άτομο αγνώστου κινδύνου, ενώ το άτομο το οποίο, για παράδειγμα, έρχεται 25η φορά στα σύνορά μας, ε, του λέμε ουσιαστικά ότι αποτελεί άγνωστο επίπεδο κινδύνου. Ποιος είναι ο σκοπός του συστήματος. Να μην θεωρείται άγνωστο κινδύνου το άτομο που έρχεται 25η φορά, για παράδειγμα, στα σύνορά μας αποτελεί αυτό διακριτική μεταχείριση. Δεν νομίζω. Αυτό τι θα σήμαινε αν θεωρούσαμε ότι αυτό είναι διακριτικό σύστημα και προκαλεί διακρίσει, ε, θα σήμαινε ότι και το σύστημα συνοριακών ελέγχων και αυτό συνεπάγεται διακριτική μεταχείριση. Γιατί επιλέγει να; μία ομάδα για ελέγχους. Ιδάλλως θα πρέπει να κάνουμε ανταλλαγές ελέγχους για όλους. Σε, σε ό,τι αφορά το τεχνικό σκέλος και το κόστος, κατανοώ τις ανησυχίες και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε από κοινού. Θα πρέπει το κόστος να εκτιμηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και προφανώς αυτοί οι υπολογισμοί θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου για να δούμε και το τι θα εγκρίνει τελικά ο συνομοθέτης και θα είναι οι που χρειάζεται να εφαρμοστούν και άρα εξορισμού θα πρέπει εκ νέου να γίνουν υπολογισμοί σε ό,τι αφορά ενδεχόμενε περικοπέ που μπορεί να προκύψουν στο επόμενο δεσυνομικό πλαίσιο. Υπάρχουν ε, επιλογές που θα πρέπει να γίνουν. Είναι πολιτική φύσεω. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τις κάνουν. Αν περιοριστεί ο σχετικό προπολογισμό, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε θα μειώσουμε τα εθνικά προγράμματα για τα κράτη-μέλη. Θα περιορίσουμε την κάλυψη του κόστους για το σύστημα ευφυών συνόρων και πάλι όμως δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση ναι ή όχι. Θεωρούμε ότι θα μπορέσει να καλυφθεί για παράδειγμα η ανάπτυξη του συστήματος το κατά πόσο θα καλυφθεί για παράδειγμα και η συντήρηση του συστήματος το πρώτο έτος είναι κάτι άλλο. Θα το δούμε. Από τεχνική άποψη θα πρέπει να εξετάσουμε μαζί με τους εμπειρογνώμονες τα συστήματα αυτά, αλλά και πάλι η βασική ιδέα είναι τα συστήματα να αναπτυχθούν βάσει τη υφιστάμενη πλατφόρμας που υπάρχουν για τα συστήματα για τις θεωρήσεις και εξορισμούς θα πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές τράπεζες δεδομένων για τα συστήματα αυτά και θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες πρόσβασης για τα συστήματα αυτά, να μην υπάρχει τέτοια περίπτωση σύγχυση. Ένα τελευταίο σημείο για το κατά πόσο θα πρέπει να προχωρήσουμε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ΕΣΤΑ, όπως υπάρχει στη ΣΥΠΑ. Έχουμε κάνει μια μελέτη για την προστιθέμενη αξία ενός τέτοιου συστήματος και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει επαρκής ε, προστιθέμενη αξία που θα μας οδηγούσε στην κατεύθυνση αυτή. Θα δούμε τι θα γίνει και με το μέλλον της πολιτικής για τις θεωρήσεις του 2014, αλλά μέχρι τότε δεν σκοπεύουμε να υποβάλουμε σχετικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μποταρέλη, επειδή σας έθεσα δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις, αν θα μπορούσατε να τις απαντήσετε είτε προφορικά είτε γραπτά σε ό,τι αφορά τις εμπειρίες των, ε, του Αμερικανικού συστήματος εισόδου-εξόδου, πώς λειτουργήσε αυτό και κατά δεύτερον από τεχνικής άποψης είναι εφικτό και επιτρέπεται στα πλαίσια των κανόνων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου να ζητηθεί από μια εταιρεία να αναπτύξει ένα τέτοιο σύστημα που δεν εντάσσεται στα πλαίσια του Patriot Act. Δεν ξέρω, θέλετε να απαντήσετε τώρα, εδώ και τώρα ή γραπτά. Um, ε, το 50%. Για την πρώτη σας ερώτηση, να εξετάσαμε προσεκτικά την εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τη μια βλέπουμε αρκετά μεγάλες διαφορές ως σημεία φετηρία Ξεκίνησαν, είπαμε, ένα σύστημα που δεν υπήρχαν έλεγχοι εξόδου σε κανένα στα σύνορα. Δηλαδή, όταν έβγαινε κάποιο από την επικρατεία του, δεν υπήρχε έλεγχο στα σύνορα και έτσι λοιπόν εξορισμού είναι πολύ πολυπλοκό να οικοδομήσει κανεί ένα σύστημα εισόδου-εξόδου. Εμεί ξεκινάμε από άλλη εφετηρία γιατί είναι υποχρεωτικό για όλε να ελέγχονται στην έξοδο συνόρων του χώρου Σέγγεν. Ξεκινάμε λοιπόν από διαφορετικές αφετηρίες και θα έλεγα ότι το σύστημα των ΙΠΑ είναι ένα πολύ μεγαλύτερο σύστημα ως προς το στόχο και το τι θέλει να πετύχει. Ενώ αυτό που προτείνουμε εμείς είναι πιο στενό και πιο συγκεκριμένο. Όμως και κάτι συγκεκριμένο σημειώσαμε τα προβλήματα που βίωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν βιομετρικά στοιχεία και αυτό είναι ένας από τους λόγους που προτείναμε το μεταβατικό στάδιο ε, για να υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος προσαρμογής. Παραδείγματο χάρη, να μην ε, πάμε στο τελευταίο στάδιο από την πρώτη μέρα, αλλά να το κάνουμε σταδιακά και να βασιστούμε στην εμπειρία που θα αποκτούμε σύν το χρόνο. Τώρα για τη δεύτερη ερώτησή σας δεν έχω ιδέα. Θα προσπαθήσω να βρω κάποιον που ξέρει και θα προσπαθήσω να επανέλθω. Ευχαριστώ κύριο Μπουταρέλη. Ευχαριστώ. Θα επικεντρωθώ στο ερώτημα της κυρίας Ζόμερ καταρχήν αλλά επίσης ε, θα αναφερθώ και μέσω στο όσα είπατε. Είπατε πότε, σύντομα είναι η απάντηση, τις επόμενες εβδομάδες. Ε, σήμερα ξεκινάει η Άνοιξη και εν τω μεταξύ είμαστε έτοιμοι για μια άτυπη συνεδρίαση με τους συζήτητες και για να μοιραστούμε μαζί σας ε, τα άτυπα σχόλια που εκδώσαμε, που δημοσίευσαμε πέρσι τον Αύγουστο και το 2008. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε το πακέτο των ευφυών συνόρων. Βεβαίως, το θέμα αυτό θα το δούμε από μια συγκεκριμένη σκοπιά, δηλαδή την προστασία των δεδομένων, που δεν είναι και τόσο ίσονο σημασία έτσι όπως φαίνεται. Επίσης, εσείς ασχολείστε και με το πολιτικό θέμα, το κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προτεραιότητες. Εξετάσουμε το κόστος όχι μόνο σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και τα ωφέλη. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας ε, δεν είναι μόνο βέλτιστε πρακτικές ή συστάσεις, αλλά είναι νομικές απαιτήσει. Οποιαδήποτε λοιπόν πρωτοβουλία είναι νόμιμη αν ε, πραγματικά σέβεται αυτό το τεστ, περνάει το τεστ της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. Δηλαδή θα εξετάσουμε το θέμα της πρόσβασης των διοικητικών οργάνων, το θέμα της αποθήκευσης ε, των δεδομένων, που θα βρίσκονται τα δεδομένα, και άλλα ζητήματα αναλογικότητας, όπως η χρήση βιομετρικών στοιχείων. Αλλά η κύρια ανησυχία μας είναι πράγματι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σύστημα για να πετύχουμε τους στόχους. Που αναφέρονται στις προτάσεις. Ναι, νόμιμη μένει στόχη αυτή. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε όσους ε, παραμένουν ε, παραπάνω παρανόμως, αλλά χρειαζόμαστε ένα τόσο μεγάλο όγκο συλλογής δεδομένων για να πετύχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Εγώ ασχολούμαι με την προστασία των δεδομένων για πάνω από 20 χρόνια, αλλά ήμουν δικαστής στο παρελθόν και ο κύριος ε, Κολλιού θα θυμάται πριν 11 χρόνια τότε ήταν ε, πρόεδρος ε, της Εποπτικής Αρχής Ένγκεν και συζητούσαμε τις τροπολογίες για το ΣΥΣ 2 που αναμενόταν να μπει σε σύντομα ε, σε λειτουργία. Και βλέπετε τι συμβαίνει 11 χρόνια αργότερα, ποιο είναι το πλαίσιο. Ανέφερα την ανάγκη να έχουμε και μια μελλοντική ένα μελλοντικό όραμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες και βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται για διάφορους σκοπούς και στόχους και πολλές φορές έχουμε επικαλύψεις. Δηλαδή, έχουμε διαφορετικές απαιτήσει, έχουμε συστήματα που επί χάρτου είναι ενδιαφέροντα, στη θεωρία ενδιαφέροντα, αλλά όχι στην πράξη. Μήπως να μιλήσουμε για τα τελωνιακά συστήματα πληροφόρηση, και δραστηριότητε που αναπτύσσονται γύρω από αυτά τα συστήματα που δεν χρησιμοποιούνται ακριβώ έτσι όπω αναμενόταν. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε και μία ανάλυση για τις προοπτικές για το μέλλον και αυτό αφορά και όλες τις πλατφόρμες σε όλους τους τομείς του πρώην τρίτου πυλώνα. Βεβαίω, οι νέε πρωτοβουλίε βασίζονται σε παρελθούσα εμπειρία και θα πρέπει να αναλύσουμε και την παρελθούσα εμπειρία όταν θα υλοποιήσουμε αυτό το εγχείρημα σε σχέση με τις ε, πρωτοβουλίες ε, που λαμβάνονται τις ορισμένα κρατημέλη και θα είμαστε τόσο δυνατόν προδραστικοί ως συνήθως, αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι τελικά δεν θα είμαστε σκεπτικοί ή επικριτικοί. Πιστεύω ότι η έμφαση έγκυται σε όσα είπε ο κύριος Τόρβαλτς Δηλαδή επικεντρωνόμαστε στους σκοπούς και γνωρίζουμε ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία και τα νούμερα. Και πάλι η κυρία Κέλλερ αναφέρθηκε ε, στο θέμα ε, των επιπτώσεων στις αρχές προστασίας του δεδομένου. Αλλά και πάλι έχετε εσείς μια ευκαιρία να κάνετε τη σωστή επιλογή. Μας βάζετε πολύ μεγάλη ευθύνη στους ώμους μας. Ωραία. Εδώ τελείωσε η συζήτηση αυτή. Ευχαριστούμε τους ομιλητάς. Μου ζήτησαν να σας υπενθυμίσω ότι συνεχίζουμε και το απόγευμα στις 3 ο κύριος Ράιτ θα έρθει για να μας μιλήσει για τα εγκλήματα.